Good, liebe... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής και πριν περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης ήθελα επί τη ευκαιρία και είναι και σχετικό με το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη να παρακαλέσω μια και θα φύγει ο Μάρτι Κάρλαος, ο αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση στην TTIP, που έχει δουλέψει χρόνια τώρα στην Επιτροπή μας, πολύ εντατικά, έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά θέματα, ιδιαίτερα μετά την συνθήκη της Λισαβόνας και τις ενισχυμένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πολλά θέματα, μεταξύ άλλων και την TTIP και την ΣΕΤΑ. Στι 15 λοιπόν του μηνό, αν δεν απατώμε, ο Μάρτιν θα φύγει, 15 Μαρτίου. Θα πάει, δεν θα πω στου αντιπάλου, αλλά στου εταίρου τη Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα μεταβεί. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευχόμαστε και για μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της δικής του παρουσίας εκεί να γίνει πιο θετική και φιλική προς το Κοινοβούλιο. Κάθε καλό λοιπόν Μάρτιν. Και τώρα πάμε στο σημείο 14, TTIP. Μετά τη συζήτηση που ξεκινήσαμε με το εγγραφό εργασία που υπογράφω εγώ και τα σχόλιά σας που συνέλεξα προσπαθώ να διατυπώσω μια πρόταση ψηφίσματος ικανή να συλλέξει την υποστήριξη της πλειονοψηφίας εδώ στην ομάδα, στην Επιτροπή μας Πρέπει να προσδιορίσουμε και το θέμα το χρονικό, το χρονοδιάγραμμα. Γιατί έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, ξέρετε. Με νέους ευρωβουλευτές κατά το ίμιση, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αποτελεί αυτό και μια ευκαιρία για μας να επαληθεύσουμε για μια φορά πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την TTIP, για την TTIP. ένα θέμα το οποίο έχει προξενήσει πολλές και επικριτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των πολιτών, τα κράτη-μέλη. Έχουν κυκλοφορήσει πολλές φήμες, έχουν εκφραστεί πολλές ανησυχίες και φυσικά για μας ως προσώπους των κρατών μελών, των πολιτών των κρατών μελών, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και τα λαμβάνουμε υπόψη. Ήταν λοιπόν κατάλληλη χρονική στιγμή εν ώψη και της δυναμικής των διαπραγματεύσεων, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι που είναι εδώ και ο Ιγνάσιο Πιζέρο, ο οποίος ανέλαβε και διεξήγαγε εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις συνομιλίες. Έχουν διεξαχθεί 8, 8 γύροι διαπραγματεύσεων αλλά νομίζω συμφωνούμε πως δεν έχουμε καταλήξει ουσιαστική συμφωνία. Αυτό ασφαλώς σχετίζεται και με το γεγονός ότι από την ε, άλλη όχθη του Ατλαντικού οι εταίροι έχουν θα έλεγα δείξει ελλειπή στάση σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε εμείς. Τώρα προχωρούμε σε βάθηση των ε, συνομιλιών και τον συστήσω εδώ στο Κοινοβούλιο. Την τρέχουσα ίσως και την επόμενη εβδομάδα ξέρουμε ότι και το ε, Κογκρέσο και η Γερουσία του Ευρωπαϊκού του, των Πολιτείων θα συζητήσουν τα θέματα και πάλι για να δώσουν στη δυνατό, στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε σύναψη της συμφωνίας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και σήμερα με ε, εκπρόσωπο του Κογκρέσου που μας λέει ότι η τελική υποβολή για έγκριση στο Κογκρέσο προβλέπεται το Μάιο. Και άρα μπορούμε να έχουμε μια παράλληλη τοποθέτηση του Αμερικανικού Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συναδελφοί, μου φαίνεται πολύ εύστοχη αυτή η παράλληλη πορεία. Ύστερα από 1,5 χρόνο συνομιλιών μεταξύ των διαμεσολαβητών, των διαπραγματευτών ήρθε η ώρα και τις δύο χθες του Ατλαντικού οι νομιμοποιημένοι και δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών να αξιολογήσουν μέχρι που έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις και που θέλουμε να δούμε πιο συγκεκριμένες πρόοδους. Εξού και το ψήφισμα που έχουμε να εξεργαστούμε. Προτείνω λοιπόν ψήφισμα επί τη βάση του άρθρου 108 παράγραφος 3η ή 4η του κανονισμού μας, όχι το συνηθισμένο δηλαδή είδος ψηφίσματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν ώστε δυνατόν περισσότερες επιτροπές στην επεξεργασία του ψηφίσματος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιληφθεί μόνο μία επιτροπή από το Κοινοβούλιο, αλλά να έχουμε στο δυνατόν ευρύτερο φάσμα ε, θέσεων και προτάσεων. Νομίζω ότι γνωμοδότηση με 14 επιτροπές δεν είχαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον σε ψήφισμα της δικής μας επιτροπής. Ο προγραμματισμός λοιπόν. Θα εξετάσουμε σήμερα το σχέδιο ψηφίσματος και θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω επεξεργασία ώστε να είναι δυνατόν η Ολομέλεια να εγκρίνει το Μάιο το ψήφισμα όπως εξήγησα παράλληλα και με την εξέταση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Στην πρότασή μου αναφέρομαι σε πέντε τμήματα, πέντε ομάδες θεμάτων. Το μεγάλο θέμα TTIP, το ευρύ θέμα TTIP καταρχάς, το οποίο έχουμε διεξοδικά συζητήσει, είχαμε και ένα ψήφισμα για την TTIP την ίδια. Και άρα τώρα αυτό που μου μένει να αιτιολογήσω γιατί θέλουμε μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να αναλάβουμε αυτές τις πραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Συμφωνία για να ε, ορίσουμε κανόνες για τις συναλλαγές με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια χωρίς κοινωνικό ή περιβαλλοντικό dumping κανόνες δηλαδή ισοδίκαιους εν ώψη της παγκοσμιοποίησης. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ ε, το 50% του παγκοσμίου ΑΕΠ ανήκει στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε ορόσημα για την παγκόσμια οικονομία. Και επίσης, εάν κοιτάξουμε και τις παγκόσμιες εμπορικές διασυνδέσεις και συναλλαγές, ασφαλώς μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μεγάλη δυνατότητα απήχησης και σταθεροποίησης των εμπορικών σχέσεων και των επιμέρους, των δηλαδή των κρατών μελών. Κατά τρόπον ώστε οι συναλλαγές αυτές να λειτουργούν προς όφελος των εργοδοτών και των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις λοιπόν, ε, τρία θέματα στις διαπραγματεύσεις. Στα οποία αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα έχουμε την πρόσβαση στις αγορές. όπου έχουμε κάθε συμφέρον να αναλάβουμε μια πιο αποφασιστική δράση, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν ε, σε πολλούς τομείς ε, αγορές κατακυρματισμένες ε, και έτσι με την εξάλληψη των δασμών ή των δασμολογικών ποσοστώσεων μπορούμε να φέρουμε κάποια βελτίωση. Αυτό ισχύει για τα βιομηχανικά, τα γεωργικά προϊόντα και άλλα. Αλλά και για τις δημόσιες συμβάσεις. Το Buy America Act, παραδείγματι, μπορεί να δώσει μια καλή ευκαιρία για πρόσβαση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Μπορούμε να λάβουμε μια δράση αποφασιστική ως εκ τούτου για τα θέματα αυτά συνολικά. Και η δεύτερη, το δεύτερο θέμα, η σώμα των διαπραγματεύσεων, πιο περίπλοκο, αφορά τα μη δασμολογικού φραγμούς στο εμπόριο. όπου μπορούμε να πούμε ότι είτε προχωρούμε σε κοινέ προδιαγραφές για αμοιβαία αναγνώριση, είτε σε αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών που θα θέλαμε να απαριθμίσουμε ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν σε πολλούς τομείς ε, δυνατότητες να γίνουν δεκτές κοινέ προδιαγραφές γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους έχουμε η μεν και η δε Ανατολική και Δυτική Όχθη του Ατλαντικού διαφορετική θεώρηση. Άρα μπορούμε να έχουμε πιθανόν λίγες κοινέ προδιαγραφές επί παραδείγματο το σύστημα πέδησης ABS για τα και σε άλλους τομείς μπορούμε να ρυθμίσουμε πολλά ζητήματα με την αμοιβαία αναγνώριση και τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση που έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί έτσι θα είναι ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προϊό, παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Πολλοί είναι οι τομείς που μπορούν να δώσουν εδώ συγκεκριμένα παραδείγματα και μόνο αν σκεφτούμε ότι θα αποφεύγεται η διπλή διαδικασία πιστοποίησης Πολύ συγκεκριμένα μια μικρομεσαία επιχείρηση ευρωπαϊκή, η οποία ούτω ή άλλω χρειάζεται την πιστοποίηση στην Ευρώπη, φερειπίν ε, για ιατρικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θα χρειάζεται, χρειάζεται προς το παρόν αντίστοιχη πιστοποίηση στι ΗΠΑ, ενώ οι διαδικασίε είναι οι ίδιες. Η λεγόμενη παραγωγή just in time, για μικρομεσαίες επιχειρήσει μπορεί να έχει πολύ καθοριστική σημασία το εάν ένα προϊόν χρειαστεί να περάσει κάποιες ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη περισσότερο χρονικό διάστημα περιμένοντας την διεκπαιρέωση των τελωνιακών διαδικασιών. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην σταθεροποίηση και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Έδειξαν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις εδώ και 1,5 χρόνο και τα θέματα στα οποία δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία αναγνώριση, ακριβώς γιατί έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις στα χημικά επιπαραδείγματα γιατί εμείς στην Ευρώπη με την ε, οδηγία, με τον κανονισμό Ρίτσι έχουμε πολύ συγκεκριμένη ε, νομοθεσία εκτεταμένη, καλύπτει τεράστιο αριθμό χημικών ουσιών επικίνδυνων για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον και αντίστοιχα προβλέπει τη διαδικασία της αδειοδότησης ή την απαγόρευση άδειας κυκλοφορίας, κάτι που δεν προβλέπεται στην δυτική όχθη του Ατλαντικού και άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε αμοιβαία αναγνώριση. Πάντως μπορούμε να εξασφαλίσουμε αμοιβαία ενημέρωση για την αξιολόγηση των κινδύνων. Στο χώρο των τροφίμων επίσης, παραγωγής τροφίμων. Με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές έχουμε νομοθεσία στην Ευρώπη πολύ διαφορετική από αυτήν των πολιτειών και εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί αμοιβαία αναγνώριση, γιατί δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μπορούμε να τα διαχειριστούμε με το σύστημα των, ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Ακούσαμε και το πρωί θέματα σχετικά και νομίζω για την τρίδα και έτσι στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων μπορούμε να δούμε με μια θετική ε, λίστα ποιες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μπορούν ε, να συμμετάσχουν στις δημόσιες, στη δημόσια παροχή υπηρεσιών ακριβώς για να διαφυλαχθεί η ποιότητά της. Η τρίτη θεματολογική ενότητα, αγαπητοί φίλοι, και πιο διαφιλονικούμενη, αυτή στην οποία θα θέλαμε στο δυνατόν πιο σαφή τοποθέτηση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμπεράσματα έχουμε αντλήσει από την εμπειρία μας μέχρι τώρα από τις διαπραγματεύσει και τι περιμένουμε για να χαρακτηρίσουμε θετική την έκβαση των διαπραγματεύσεων έχει να κάνει με την γεωγραφική, για το γεωγραφικό προσδορισμό προελεύσεως που θέλουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε να εφαρμόσουν. Θέλουμε λοιπόν γεωργικά προϊόντα ευρωπαϊκά να είναι δυνατόν να προστατεύονται με τους ίδιους όρους και στις ΗΠΑ και η παραγωγή ε, περιφερειακής εμβέλειας να ε, προστατευθούν όταν τα προϊόντα τους κυκλοφορούν στις ΗΠΑ με κανόνες αντίστοιχους, με κανόνες που θα εξασφαλίσουν και δυνατότητες συνεργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Και έτσι θα εστιαστούμε σε ένα κοινό σώμα κανόνων και προδιαγραφών που θα χρειαστεί περαιτέρω να επεξεργαστούμε, χωρίς βέβαια αυτό να θέτει ένα αμφιβόλο τις δημοκρατικές διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων που έχουμε. Μέχρι τώρα οι προτάσεις για τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν με έχουν επίση και έτσι η ρυθμιστική συνεργασία όπως ονομάζεται ε, βλέπουμε ότι δεν επιτρέπει την εμπλοκή των ε, ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, αλλά τον προσδορισμό από τις ρυθμιστικές λεγόμενες αρχές. Τώρα ή θα πρόκειται για προδιαγραφές ίζο η ομάδα εργασίας του 20, ε, το 29 ε, της Γενέβης θα δούμε πώς διαμορφώνονται αυτές οι προτάσεις. Πάντως θέλουμε να έχουμε προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την καθοριστική απόφαση από πλευρά του Δημοκρατικά Εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προστασία των επενδύσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολλούς, έχει μεγάλη σημασία. Σημειώνεται σημαντική εξέλιξη ως προς την τοποθέτησή μας και νομίζω ότι μπορούμε να προστατεύουμε τους επενδυτές εφόσον μπορούμε και να βλέπουμε σωστά το καθήκον, το έργο το οποίο επιτελούν με βάση και τις, με τις κατευθύνες του ΩΣΑ. ώστε να μην υφίσταται οι δικοί μας επενδυτές αρνητικές διακρίσεις. Αντίστοιχα όμως δεν θέλουμε και να ε, βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση οι άλλοι επενδυτές. Θέλουμε μια ισότιμη μεταχείριση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και την αναζήτηση μιας δικής λύσης σε προβλήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Ο, τρί, ο τέταρτος τομέας θεμάτων που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα έχει να κάνει και με το γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτή την σύμβαση για τις εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή το προσδιορισμό ε, προδιαγραφών και να κάνουμε ως εκ τούτου ανταγωνισμό με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας και όχι με όρους dumping. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο βιωσιμότητας με προδιαγραφές όμως που θα καλύπτουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλογιστούμε το πώς ε, συμπεριφέρονται αλλοδαπές ε, επιχειρήσεις που δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα ευρωπαϊκές στις ΗΠΑ αλλά και άλλο. Θα πρέπει οι να ισχύουν πάντοτε. Και ένα ακόμα, μια ακόμη θεματική ενότητα που αφορά την ε, διαφάνεια και την συνεργασία. Είμαι πεπισμένος, ακράδαντα, ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα αυτό θα το επιτύχουμε μόνο εφόσον έχουμε στο δυνατόν ε, ευρεία και ειλικρινή συζήτηση με όρους διαφάνειας και με εξασφάλιση τη διαφάνεια αυτή όχι μόνο για τους βουλευτές αλλά και για την κοινή γνώμη. Αυτά λοιπόν οι δικές μου θέσεις και περιμένω με αδημονία να ακούσω τα σχόλιά σας. Ο, κύριο κύριος Κάσπαρη εκπροσωπεί την κυρία Κουίστολ Τρόβολτ και λαμβάνει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ. η συνάδελφο δυστυχώ ε, ασθενεί αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό με παρακάλεσε να ζητήσω εκ μέρου τη συγγνώμη και να σα απευθύνω του χαιρετισμού τη. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την καλή έκθεση. Η προσέγγιση είναι ήδη σαφής πιστεύουμε στο σημείο 1αε, ότι δηλαδή πρέπει να καταστεί η TTIP μια συμφωνία για τη διαπραγμάτευση με όρους διαφάνειας, μια συμφωνία η οποία θα ενισχύει τον ανταγωνισμό σε όρους υγιής και θα βοηθά στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Θα ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα εξασφαλίζει δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, για δράση χωρίς να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Τώρα, ζήτημα θα είναι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει και την πλειονότητα των συναδέλφων εδώ στο Κοινοβούλιο Θέλουμε την TTIP μεν, αλλά όχι πάση θυσία δε. Δεν θέλουμε δηλαδή να κανουμε αρονάρον μια διαστική δουλειά. Θέλουμε η ευκαιρία που έχουμε να αξιοποιηθεί, να αξιοποιήσουμε για το συμφέρον των πολιτών μας την ευκαιρία αυτή για σωστές και ομαλές διαπραγματεύσεις, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Είναι καλή η πρότασή σας, αποτελεί μια πρώτη καλή προσέγγιση στη νέα αυτή θητεία μας και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει και μας αρέσει το ύφος της εκθέσεως. Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην βρέψουμε το σφάλμα, να, ορίσουμε, να διατυπώσουμε όρους ή προϋποθέσεις, γιατί ξέρουμε ότι η Επιτροπή είναι εκείνη η οποία διαπραγματεύεται. Τον Μάιο του 2013 με μεγάλη πλειονοψηφία με την έκθεση ΟΡΕΒΑ ε, εγκρίναμε ένα ψήφισμα το οποίο βλέπουμε να επανέρχεται σε όρους και πιο λεπτομερείς στη δική σας πρόταση. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ευρύτατη συνένεση. Για τη ρυθμιστική συνεργασία θα χρειαστεί να δουλέψουμε πολύ εντατικά, αλλά πρέπει να αποτελέσει κομμάτι της TTIP. Στη διαφάνεια πρέπει να δούμε περισσότερες προόδους. Με τη νέα Επιτροπή και κυρίως με την Επίτροπο Μάλστρομ μπορούμε να περιμένουμε καλύτερες, ε, καλύτερα ακόμα υποτελέσματα από τόσο έχουμε μέχρι τώρα δει. Στη διαφάνεια πάντως που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ ως Κοινοβούλιο θέλουμε να τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες και να μην δούμε συνέπειες διαπραγματεύσεων ε, οι οποίες θα αποβούν ίσως και ε, δυσμενείς για τους πολίτες μας. Πάντως πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλή. Έχουμε τις τροπολογίες μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τις νομοδοτήσεις των λοιπόν επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου με τις προτάσεις για τροποποίηση, συμπλήρωση. Η αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να βγει πλέον από την ε, σκιά η, εμπορική, η διεθνής εμπορική μας πολιτική, όπου βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό, ε, νομίζω ότι είναι μια δουλειά που έχει γίνει έστω και χωρίς πολύ μεγάλη προσοχή από την, από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Έχουμε κάνει μια πολλή δουλειά ε, τα τελευταία χρόνια είτε για τη σχέση με την Κορέα είτε για τη σχέση με το Περού. Νομίζω ότι βλέπουμε πως για τα ζητήματα των ελάχιστων εγγυημένων δημόσιων υπηρεσιών και άλλα πολλά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει δουλειά αξιόλογη, αξιόπιστη, έχουν αναλάβει έμπειρα και ικανά χέρια να επεξεργαστούν τα θέματα αυτά και γι' αυτό χαιρόμαστε με, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει προοπτική για περαιτέρω καλή και επικοδομητική συνεργασία με αποτέλεσμα τελικό την TTIP όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Μια TTIP την οποία θα μπορούσε να υπερψηφίσει ε, με συντριπτικές πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, Κέμπλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάκιν επίσης ε, κλινήρισε δυστυχώς ε, και μιλάω εγώ εξ ονοματό του. Είμαστε σε σημαντικό σταυροδρόμι σήμερα για την TTIP. Ε, και καλωσορίζουμε αυτόν τον απολογισμό πολιτικής κοφιάς όπως μας πρότεινε και ο Πρόεδρος όμως ε, είμαστε σχετικά πρόωρα στάδια της διαπραγμάτευσης ε, δεν υπάρχει ακόμη κοινό κείμενο και το να ορίζουμε εμείς τις κόκκινες γραμμές μας ενώ δεν υπάρχει τίποτα επιτάπητος είναι πρόωρο και μπορεί να αποβεί και αντιπαραγωγικό. Ευχαριστώ τον εισηγητή πάντως γιατί είναι λογικό στην προσέγγιση που υιοθέτησε στο μέτρο που δεν απέσυρε τίποτα. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία και θα επανέλθω σε αυτόν αυτό το χρόνο. Παρόλα αυτά με ιδιαίτερη προσοχή φροντίσατε να μην αποκλείσετε τίποτα και το εκτιμούμε αυτό. Ε, πρόκειται και για να μείνουμε προ του Αμερικανούς εταίρους μας, διότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και δεν μπορούμε να ζητούμε πράγματα ενώ οι ίδιοι δεν έχουμε εξετάσει όλες τι εναλλακτικέ λύσεις. Για τι ε, λεπτομέρειε ε, μέσα στα εκτιμώντα, μιλάτε για τον τη σημασία, για την προστασία των καταναλωτών, Φυσικά αληθεύει αυτό. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη η πλειοψηφία υποστηρίζει μια τέτοια εμπορική συμφωνία ΕΕ ε, και ε, έρευνες δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από τα 2 τρίτα, δηλαδή 65% ε, του ε, κοινού υποστηρίζει την ε, TTIP. Στη Λουθανία το ποσοστό φτάνει και το 80-90%. Μόνο σε δύο κράτη-μέλη υπάρχει πλειοψηφία κατά της συμφωνίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ευσταθεί λοιπόν ότι δεν επιθυμούν να συναυθεί αυτή η συμφωνία οι πολίτε. <clears throat> Φυσικά είναι πιο σημαντικό το περιεχόμενο σε σχέση με την ταχύτητα, αλλά θα πρέπει να συμφωνηθεί το πακέτο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια καταρχάς συμφωνία και να επανέλθουμε στη συνέχεια. Όμως μια πλήρη συμφωνία είναι ε, ο μοναδικός τρόπος, μονόδρομος, ε, διότι αλλιώς ε, αν βιαστούμε θα δείξουμε ότι δεν είμαστε και φιλόδοξοι. Ε, τώρα πώς επηρεάζονται τα παγκόσμια πρότυπα. Ε, είναι σημαντική ευκαιρία που μας δίνεται. Είπαν εξάλλου πολλοί ότι αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΕ δεν καταφέρουν να συνάψουν τη συμφωνία, τι συνεπάγεται αυτό για μελλοντικέ συμφωνίες με την Ινδία, την Κίνα, πολύ σημαντικές οικονομίες με τις οποίες φαντάζομαι θα έχουμε πολύ σοβαρότερα προσκόμματα για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών σε σχέση με τη των αναλογιών είναι πιο εύκολα τα πράγματα με την TTIP. Για το θετικό κατάλογο τώρα και τη σχετική προσέγγιση για τις εταιρείε. δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετά φιλόδοξη η πρόταση. Προτιμούμε τον αρνητικό κατάλογο, αλλά στην καλύτερη περίπτωση θέλουμε να έχουμε ένα μεικτό σύστημα καταλόγων, ούτω ώστε να μην χρειάζεται να περάσουν όλοι από τι υπηρεσίε για να έχουν πρόσβαση στο θετικό κατάλογο. Με το μεικτό ε, σύστημα ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε άλλου του εισαγωγικά μεσα ε, Κάτι που παραμένει ασαφές για πολλούς είναι οι δημόσιες υπηρεσίες εξαιρούνται από την ε, συμφωνία και αυτό βοηθάει όμως θα θέλαμε οι διαπραγματευτέ να κάνουν σαφή ρητή δήλωση ε, ε, όπου αποκλείουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να ε, αναφερθεί αυτό ρητό. οι βασικοί διαπραγματευτές είπαν ότι υποστηρίζουν μια τέτοια ιδέα και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει αυτό και θα σταματήσει η συζήτηση για τις δημόσιες υπηρεσίε υπηρεσίες μία και έξω. Για το ISTS γιατί προστασίας επενδυτού, ε, σε σχέση επενδυτή κράτους. Δεν αναφερόμαστε, δεν αναφέρεστε κύριε Σιγητά σε συγκεκριμένο σύστημα, μιλάτε για απουσία διακριτικής μεταχείρισης κατά των επενδυτών. Πρώτον, περάσουμε τώρα στο να μιλάμε για ε, εκπόνηση νομικών συστημάτων, Εκφράζεται την άποψή σας ότι δεν επιθυμείτε να κατοχυρωθεί ένα σύστημα ISDS. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε. Ε, υπάρχουν χώρες όπως οι δικές μας όπου υπάρχει ένα σχετικό νομικό σύστημα και ε, σε, στα πλαίσια όμως διεθνών συμφωνιών δεν σημαίνει αυτό ότι εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις. Ε, αντιπροτείνεται ένα μηχανισμό state to state από κράτος σε κράτος. Όμως αυτό να έχει παγίδες, ε, μπορεί να αποκτήσουν κάποια στιγμότα πολιτικές διαστάσεις και αυτό αντιβαίνει στο στόχο σας να καταργήσουμε την διακριτική μεταχείριση και ένα άλλο μειονέκτημα με αυτό το σύστημα είναι ότι δεν θα εξεταστεί Ενδεχομένω σε μία περίπτωση επιχείρησης, διότι μπορεί να κρίνει ένα κράτο ότι για διπλωματικούς, για πολιτικούς λόγου δεν θα πρέπει ε, καν να εξεταστεί το ζήτημα παρά το, τη ζημιά που θα έχει υποστεί η επιχείρηση. Λοιπόν, συνοψίζοντας, ε, ε, θεωρούμε ότι στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι η συμφωνία TTIP αντί να λύσει τα προβλήματα που πρέπει να λύσει. Το ISTS, αυτό το σύστημα διευθέτης διαφορών επενδυτή κράτους δεν είναι κάτι καινούριο, δεν εμφανίστηκε τώρα με την TTIP. Ε, ε, Υπάρχει από τη δεκαετία του 70 και δίνει τη δυνατότητα οι πολυεθνικές να ε, καταθέσουν, ε, μπορούν να καταθέτουν αγωγές ε, κατά των κρατών λέτε εσείς, και να διεκδικούν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί έχουν γίνει σχετικές μελέτες και εξάλλου δεν αναφέρεται ότι μπορεί και να χρειαστούν ευρωπαϊκές επιχείρησεις προστασία μέσω του συστήματος ISDS. Δεν ισχυρίζομαι φυσικά ότι είναι τέλειο το σύστημα στη μορφή που υπάρχει σήμερα και όντως την έλλειψη της διαφάνειας και άλλα παρεμφερή ζητήματα ή τη μελλοντική συμπερίληψη ενός ε, ε, μηχανισμού που θα διευθετεί αυτά τα ζητήματα και μια μεταγενέστερη θεώρηση αυτού του συστήματος θα ήταν απαραίτητο, αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε διότι είναι δομικός λήθος των διαπραγματεύσεων στα μάτια των Αμερικανών και περιμένουμε τη, με του της διαπραγματεύσεως στους επόμενους μήνες με διαφορετικό έτσι ρόλο θα μιλήσω Είχαμε δέκα συναντήσεις σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο για το TTIP, το οποίο δείχνει τη σημασία αυτής της συζήτησης και χαίρομαι που το ψήσιμο αυτό έτσι μας επιτρέπει να διοχετεύσουμε, να καθοδηγήσουμε κάποιους τομείς στις επιτροπές, ώστε να δούμε ακριβώ που βρισκόμαστε σε αυτές τις σημαντικές διπραγματεύσεις. Κοίταξα στο το προσχέδιό σας, έχω αρκετά θετικά να πω όμως να πω επίσης ότι είναι κάπως διστακτικό. Νομίζω ότι ακριβώς τώρα είναι η στιγμή να εκφράσουμε την φιλοδοξία μας για μια λειτουργική και καλή TTIP. Κάποιοι λένε ίσως όχι, αλλά βλέπω ότι αυτό που κάνουμε εμείς αντανακλά τις επιθυμίες και τις ανησυχίες μας, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Πράγματι οι διαπραγματεύσεις ε, μόλις ξεκίνησαν εμείς θέλουμε να δούμε πιο απτά αποτελέσματα ώστε να καταλάβουμε που κατευθύνονται. Βλέπουμε δυστυχώς ότι η Αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται πολύ στις συμφωνίες με τις χώρες της Ασίας και έχει έτσι πολιτική καθοδήγηση σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να δούμε προς το που πηγαίνουμε και το ψήφισμα αυτό μπορεί να αποτελέσει ακριβώς ένα βήμα προς μια καλή τύπη. Φιλοδοξία μας είναι να ολοκληρώσουμε μια περιεκτική συμφωνία εμπορική και εταιρική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθεί ως υποστήριξη από την Κομισιόν από όλες τις χώρες μέλη. Μετά την εντολή είχαμε διάφορες ε, συζητήσεις με πολλούς εμπλεκόμενους, πολίτες, πλατφόρμες που δημιουργήσαμε εδώ, πάνελ, εκδηλώσεις, συζητήσεις, ΜΚΟ, think tank οργανώσεις. Μιλήσαμε σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες άτομα που προσωπούν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, ομάδες συμφερόντων και κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε τι πετύχαμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση από την Κομισιόν για διαφάνεια. Αυτή ήταν ξεκάθαρη επιθυμία του σώματος μας και χαίρομαι που έχει βελτιωθεί. Επίση χαίρομαι που το προσχέδιο αναφέρεται στο πολυμερές σύστημα. Καμιά φορά ξεχνάμε ακριβώ τη σημασία των πολυμερών συμφωνιών επικεντρωμένη στην TOTIP. Πρέπει να υπάρχει επίση και για εμά η δυνατότητα να διατηρήσουμε τον έλεγχο τη ποικιλότητα εδώ στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχει σύγχυση Επίσης, τονίσαμε τη σημασία των υψηλών προδιαγραφών, τα standards, και χαίρομαι που η Κομισιόν έκανε σοβαρές δεσμεύσει για το θέμα αυτό. Αυτό που μου λείπει όμως κάπως είναι έτσι η διεθνή συνιστόσα, δηλαδή το διεθνές πλαίσιο όπου λαμβάνουν χώρο σε αυτές τις συζητήσεις. Μπορεί στην Ευρώπη να θεωρούμε ότι έχουμε τις ψηλότερες προδιαγραφές και νομίζουν πολλοί ότι το κοτόπουλο με χλωρί είναι πολύ πιο ανθυγινό από το κοτόπουλο με αντιβιωτικά, αλλά υπάρχουν φόβοι εδώ και στην Ευρώπη για τα δικά μα πράγματα. Και αν δούμε ακριβώ τι φόβοι υπάρχουν παγκοσμίω και δεν την ποιότητα ζωή και εδώ στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με πάρα πολλού δείκτε για ευκαιρία, για ευημερία, για πρόσβαση στι δημόσιε υπηρεσίε, ε, στην εκπαίδευση, περιβαλλοντικές περιγραφές μπορούμε να πούμε ότι παγκοσμίω έχουμε ψηλότερες περιγραφές και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε όπου μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες μας οι οποίες σε σχετικούς όρου υποχωρούν γιατί ξέρετε ότι ο πληθυσμό παρουσιάζει γύρανση ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου ο πληθυσμός αυξάνεται και υπάρχουν πολύ περισσότεροι νέοι είναι λοιπόν επίγον και θα πρέπει να το τονίζει αυτό το ψήφισμα τούτο την ανάγκη για παγκόσμιες υψηλές προδιαγραφές στο εμπόριο. Αναφέρει επίσης το προσχέδιο τις προσδοκίες για το κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό επειδή είναι η αρχοκοκαλιά μικρομεσαίες της, της οικονομίας μας και υπάρχουν περιττή φραγμή για αυτές τις επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να επεκταθούν στις αγορές πέραν του Ατλαντικού. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε ότι θέλουμε αυτό το κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες να είναι φιλόδοξο. Δεν αρκεί να περιλαμβάνεται απλά και μόνο και θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα οι πιθανότητες και οι δυνατότητες εξαγωγής για τις μεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα που υπάρχει δυνατότητα δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το ότι υπάρχει περιθώριο ρυθμιστική συνεργασία για το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι υπάρχουν φόβοι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν βλέπω σημάδια από τους συναδέλφους να επιθυμούν δηλαδή μείωση ή υποχώρηση εδώ, γιατί όλοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως παίκτες και πρωταγωνιστές στη θέσπιση κανόνων και στην επίδευξη ισορροπιών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ως αποτέλεσμα της καλύτερης ρυθμιστική συνεργασία να αποφύγουμε το ενδομιλικό εμπόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η μεταφορά εξαρτημάτων προϊόντων επειδή θα πρέπει να δοκιμαστούν αποτελεί ε, έτσι, για το περιττό είναι κακό για το περιβάλλον και κοστίζει. Δημόσιοι διαγωνισμοί και πρόσβαση στι αγορέ. Μιλάτε για ισορροπία. Η ισορροπία είναι μια ήπια έκφραση όσον αφορά τι φιλοδοξίε μα. Εμεί θέλουμε περισσότερη πρόσβαση στι αγορέ, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Δεν έχει νόημα να είναι κλειστή και προστατευτική η Αμερικανική αγορά. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στη διατύπωση. Αυτό επιθυμούμε και θέλουμε να υπάρχουν μεγάλε ευκαιρίε για τι μικρέ και μεσαίε ευρωπαϊκές επιχειρήσει σε διάφορου τομεί όπω μεταφορές κλπ. Εκεί πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Επίση θέλω να δούμε τι γίνεται με τον αντίκτυπο σε τρίτε χώρε. Έχουμε μια τελωνιακή ένωση με την Τουρκία, τι γίνεται εκεί, ποιο είναι ο αντίκτυπο και το ίδιο ισχύει για το Μεξικό. Τώρα, έχω ένα ερώτημα. Το επίμαχο ζήτημα του SDS. Λέτε στην πρότασή σα ότι δεν είναι απαραίτητο να περιλάβουμε το SDS στο TTIP. Έχω ερωτηματικά. για τη ρύθμιση διαφορά μεταξύ κρατών. Για δύο λόγους. Καταρχάς, στον ΠΟΕ δεν περιλαμβάνονται επενδύσει σε αυτούς τους ε, μηχανισμούς ε, διατησίας, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικό να ζητάμε από τις κυβερνήσει να υιοθετήσουν, ας πούμε, την υπόθεση μιας ε, μικρομεσαία επιχείρησης διπλωματική σχέση με τρίτες χώρε. Ποιο καθορίζει ότι θα υπάρχει συμμεταχείριση, ποιο καθορίζει ότι θα υπάρξει λύση. Μπορούμε απλά και μόνο να εξαρτώμαστε από την βούληση της κάθε κυβέρνησης να λύνει θέματα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό αποτελεσματικό. Και μόνο χθε είδαμε προτάσεις από το πολιτικό σας κόμμα για ένα μόνιμο δικαστήριο διαιτησίας. Ωραία, το έχουμε συζητήσει αυτό. Ως μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη λύση. Αυτό όμως που προτείνετε τώρα είναι η πρόταση που θέλετε να μας υποβάλλετε γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί πολύ καιρό και πολλές διαπραγματεύσεις διπλωματικές και πολλά χρήματα για να προχωρήσει αυτό. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τι είδο συμφωνίας θα διέπει αυτό το δικαστήριο. Δηλαδή, τι είδο συμφωνίε θα θέλατε να περιληφθούν στο TOTIP, ώστε αυτές οι υποθέσεις ε, να μπορούν να πάνε στο δικαστήριο και να αποφανθεί αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτές τις τόσο επίμαχες και έντονες συζητήσεις που έχουμε θα πρέπει να έχουμε τις, τις πληροφορίες αυτές στη διάθεσή μας. Να επιθυμίσω σε όλους μας επίσης ότι είναι καλό να υπάρχει τελικά ένα καλό TTIP και ότι οι φιλοδοξίες μας δεν πρέπει να ξεπερνούν την ουσία. Νομίζω ότι το ψήφισμα αυτό παρέχει μια θαυμάσια ευκαιρία για όλους να αναφέρουν την, να μιλήσουμε τη φωνή τους ε, και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για την υποβολή της εκθέσεως καταρχάς, η οποία καλύπτει τις διάφορες πτυχές που έχουμε συζητήσει εδώ και 1,5 χρόνο στο θέμα της TTIP, περίπλοκο, πολύ σχηδές και ασαφές ακόμη όπως είναι Όλες οι πτυχές αυτές καταγράφονται στην έκθεσή σας. Εμείς λοιπόν, ως Κοινοβούλιο, αποφασίσαμε να τοποθετηθούμε σε σχέση με την επανεκκίνηση όπως ονομάσανε η Επιτροπή και η Αμερικανική πλευρά των διαπραγματεύσεων και κοιτάω να δω πού βρίσκεται η επανεκκίνηση. Διότι δεν έχει αλλάξει εντολή για τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, διότι δεν βλέπω να λαμβάνονται υπόψη τα βάσιμα μελήματα, ερωτηματικά, ανησυχίες της κοινή γνώμης, της κοινωνίας των πολιτών, των καταναλωτών. όπως θα έπρεπε. Δεύτερο, η Μαρίτσα Σάκη το έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχει αυτή η παγκόσμια διάσταση τόσο καθαρά στην έκθεση. Η Χίλαρη Κλίντον το 2011 και μετά την, από, την ε, πράξη, την νομοθετική πράξη για την ανάπτυξη της εργασίας μίλησε για μια έννοια χώρου του ΝΑΤΟ. Ε, ωστόσο αυτό χάθηκε από το διάλογο. Παραμένει όμως αζήτημα ζήτημα. Πώς παραμένουμε σε, με νέες προδιαγραφές, με νέες αρχές, κατηγορίες, ικανοί να διαπραγματευτούμε σε επίπεδο παγκόσμιου εμπορίου. Αυτή λοιπόν η σειρά αξιών και θέσεων μας που περιέγραψε τόσο καλά η Μαρίτια είναι μια, ένα σύνολο αξιών που εδώ και δεκαετίες, για να μην πω εκατονταετίες, χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας, τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία μας, η κατανάλωση, εις βάρος άλλων. Πώς λοιπόν σε μια παγκόσμια οικονομία που έχουμε διάφορους συμμετέχοντες διαφορετικούς θέλουμε εμείς να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία η οποία δεν θα επιτρέπει στους πάντες να έχουν επαρκή κατανάλωση για να εξασφαλίζουν την καθημερινή τους επιβίωση. Αυτή η πτυχή πρέπει να υπογραφμιστεί ιδιαίτερα στη συζήτηση για το TTIP. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολλά τα ερωτηματικά σε σχέση με το TTIP. Ευτυχώ, χάρη και στι πιέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ακόμη περισσότερο τη κοινή γνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε την διαπραγματευτική ε, ε, της τακτική, την στάση της απέναντι στο κοινό, αφήνει ανοιχτά τα θέματα, αφήνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει τις παρατηρήσεις του, να δει τα θέματα πιο συγκεκριμένα. Αλλά πάλι διαρωτώ με εάν θα υπάρξει κάτι καινούριο και διαφορετικό ή αν θα είναι η απόφαση που θα ληφθεί εν τέλει μόνο μερίς και μόνο εις όφελος των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και σηματοπιστωτικών οργανισμών. Εξού και το ερώτημα για τις κόκκινες γραμμές. Έχει συμφωνήσει μια κόκκινη γραμμή το Κοινοβούλιο, ο τομέας, στον τομέα του πολιτισμού συγκεκριμένα και δι των οπτικοακουστικών, όχι ολόκληρου του, του πολιτιστικού τομέα. Μένουν εκτός όμως τα, οπτικοακουστικά. Βλέπουμε όμως ότι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού πάλι έρχονται θέματα οπτικοακουστικών μέσων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσω άλλων ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, ότι θέλουμε να δυνατόν πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σαφή διατύπωση Θέλουμε να είναι ορατό αυτό το οποίο ζητούμε και σαφής η διατύπωση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τα δημόσια αγαθά, Μπέρντ, θα συμφωνήσω μαζί σου εκεί που λες ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Όμως κάνεις λόγο για αναλογικές και μετρημένες εξαιρέσεις για λογικές υπηρεσίες που θα επιτρέπουν επαρκές πεδίο διαπραγμάτευσης για τις εθνικές και τοπικές αρχές. Λοιπόν, καταλαβαίνω πού θες να το πας. Πού θέλουμε να το πάμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως. Αλλά θέλω να είμαστε πιο σοφείς στη διατύπωση. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι εδώ πρέπει να ορίσουμε σαφή ε, και μετρήσιμα ορόσημα δείκτες και να πούμε ποια είναι τα ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σχέση με την πρόοδο σε μια διατλαντική αγορά με τους Αμερικανούς η Επιτροπή αλλά και οι Αμερικανοί χρόνια τώρα μας λένε «Α, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί το κοινοτικό κεκτημένο κτλ». Μπορώ να είμαι αισιόδοξο μεν. Διότι το ζήτημα δεν είναι το πώς κινείται κανείς στην πραγματεύση, αλλά το πώς θα διαφυλαχθούν οι φυστάμενες αγορές. Και άρα σε αυτό χρειάζεται η ρυθμιστική λειτουργία, σε αυτό χρειάζεται η προσεκτική μελέτη των όρων. Και για να μην μακρηγορώ, θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με τις τροπολογίες μας στο ψήφισμα προς το όφελος των πολιτών στο σύνολό τους προς το στόχο μιας υψηλού επίπεδου ε, προστασίας για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά, για τους πολίτες προς το στόχο του, της ρητής αναφοράς των δεσμεύσεων με τι τροπολογισμού μας όπως έλεγα και μετά θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί η τελική θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, το πρόβλημα που έχουμε είναι το εξή ότι προβλέπετε μόνο ε, μία ώρα για τη συζήτηση. Άφησα του τους και ηγητές να μιλήσουν λίγο περισσότερο. Το άλλο μου δε πρόβλημα είναι ότι στι 4 έχουμε προβλέψει με την Επιτροπή Βιομηχανία στην μια ακρόαση πάλι για την TTIP. Άρα μας μένουν 8 λεπτά. για νίκη. Αγαπητέ Μπέντε, ε, δεν μπορεί να υπάρχουν προβλήματα πριν αρχίσω εγώ να μιλώ. Μετά μπορεί. Πριν όχι. Γι' αυτό το ψήφισμα ε, πολλά είναι τα θετικά ε, στοιχεία, καλογραμμένα. Με τις διευκρινήσεις που είχαμε και σήμερα το πρωί για τις δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή την ανάγκη να αναφέρουμε με σαφή τρόπο τι εννοούμε με την εξαίρεση των δημοσίων υπηρεσιών. Μπορούμε να το ενισχύσουμε την το κείμενο, αλλά νομίζω ότι σαφέστατα αναφερόμαστε πλέον στον αποκλεισμό ε, αυτών των υπηρεσιών. Πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα για τον αρνητικό και το θετικό κατάλογο. Βλέπουμε ποιοι κινδυνοι αλοχεύουν με τον αρνητικό κατάλογο ήδη σήμερα. Ο στόχος είναι να είναι κλειστός ο μηχανισμός και να περιοριστεί η δυνατότητα των κρατών να ε, κρατούν για εκείνα κάποιες υπηρεσίες, κάποιες τομείς όπου δεν θέλουν να είναι υπερβολική η Όμως όταν μιλάμε για μεικτό σύστημα με πολλούς ε, αρνητικούς καταλόγους και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να μειώσουν σημαντικά τον κατάλογο των υπηρεσιών που θέλουν να αποκλείσουν από την απελευθέρωση. Βλέπουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύστημα του αρνητικού καταλόγου Λοιπόν, θα συμφωνήσω επίσης ότι με την TTIP θα ενισχυθεί η εταιρική μας σχέση και η παγκοσμιοποίηση θα γίνει με αγαστό τρόπο και θα έχουμε ειρήνη και ευτυχία για όλους, όμως ε, δεν ασχολούμαστε καθόλου και με το, το, το βασικό πρόβλημα ε, το, τις κλιματικές αλλαγές. Ε, εξάλλου το αναφέρεις και εσύ στην έκθεσή σου ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το σχιστολιθικό. Ε, να αποκτήσουμε και εμείς πρόσβαση. Μιλάμε για την, το να αναδειχθούν τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας σε παγκόσμιο πρότυπο. Όχι, αφού δεν έχουν καν υπογράψει η ΕΠΑ. Είναι ο στόχος μας να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους. Όχι, εφόσον μιλάμε για αναθεώρηση της νομοθεσίας Dodd Frank, όχι. Λοιπόν, ο στόχος δεν είναι να επιτύχουμε πρότυπα που μας επιτρέπουν αφενός να εξέλθουμε από την κρίση και αφετέρου σε πολυμερές επίπεδο να έχουμε τις ψηλότερες δυνατές φιλοδοξίες. Δεν είναι αυτός ο στόχος όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Επίσης, ε, ως προς τη διαφάνεια, ακόμη και στα ε, εκτιμώντας, βλέπουμε ότι η μνήμα ε, αποσιάζει για την διαμεσολαβήτρια και είναι πολύ σημαντικός ο θεσμός. Ε, έχει εξασφαλίσει πολλά πράγματα για την πρόσβαση τα έγγραφα και θα καταθέσουμε τροπολογία για να αναφερθούμε στην Ευρωπαία ε, Διαμεσολαβήτρια και να αναφέρουμε ε, το γεγονός ότι ε, εάν επιθυμούμε οι μελέτες, η ανάλυση για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να γίνονται με διαφανή τρόπο θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Τώρα, σήμερα ξέρουμε πως ότι ε, θα έχουμε στις ΕΙΠΑ ε, αντιρρήσεις από πλευράς των ομόσπονδων ε, κρατών και σε εμά από τις διάφορες περιοχές σε σχέση με τον αντίκτυπο του παγκοσμίου εμπορίου και έχουμε αυτό το φόρουμ ε, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να επιληφθεί της όλης ε, ρυθμιστικής ε, διαδικασίας. Συγγνώμη, πρόκειται για ρήξη σε σχέση με την διαδικασία λήψη αποφάσεων το ίδιο το σύστημα θα αποφασίσει ποιε θα είναι οι νομοθεσίε μα για την υγεία, για το περιβάλλον, για τα κοινωνικά ζητήματα, για τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία για το καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να ενισχυθεί το, το σύστημα. Περιμένουμε και την γνωμοδότηση τώρα τη Άγκρη για τα γεωργικά ζητήματα, όμω θα έλεγα ότι για την πρόσβαση στην αγορά και για την κατάργηση των δασμολογικών ποσοστώσεων είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα που δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το γεωργικό ζήτημα μόνο με αναφερόμενοι ε, στα φυτογειονομικά πρότυπα και στην επιστημιστική ασφάλεια. Δεν ανπαρκεί αυτό. Για το ISDS θα πρέπει να αποφασίσει επιτέλους το Κοινοβούλιο. Δεν πιστεύω ε, και ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε σε μια κακή συμβαστική λύση για το ESG, γιατί είναι θέμα αρχής. Δεχόμαστε ένα νομικό, ε, δικαστικό, υπερεθνικό σύστημα ιδιωτικού δικαίου που θα υπερτερεί σε σχέση με τα εθνικά συστήματα ή με το, ε, την ευρωπαϊκή ακόμη ένωμη τάξη. λένε κάποιοι ότι με αν βελτιωθεί μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί είναι θέμα δικαιοδοσίας. Θα, ε, ούτως ή άλλως ε, ε, θα ρηθεί ο κύβος στην ψηφοφορία. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πούμε σε ένα ψήφισμα αν δεν είναι καλό το σύστημα, αλλά άμα βελτιωθεί βλέπουμε» κτλ. Όχι, θέλω να αποκλειθεί, διότι αν το γράψουμε αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να παραμείνει στην υφιστάμενη μορφή του αυτός ο μηχανισμός. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχει υπερεθνική ειδικό ε, σύστημα ε, δικαιοδοσίας, διαιτησίας, ε, λοιπόν, αυτά. Εν κατακλείδη να πω ότι υπάρχουν πολλά καλογραμμένα θετικά σημεία, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όσοι έχουν εκφράσει την άποψή του θα είναι ξεκάθαροι. Οι οργανώσεις καταναλωτών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, κάποιες εργοδοτικές ενώσεις έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε σχέση με του διαπραγματέ. Δεν μπορεί εμεί να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να καταλήξει σε κακή συμβαστική λύση. Ευχαριστούμε, κύριε Μπιγκίν. Ευχαριστώ. Κύριε Σεγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα με ενδιαφέρον το σχέδιο του Σιγητή. και εγώ ξεπλάγει που πρέπει να τον ευχαριστήσω για το ότι ένα κείμενο που συμμερίζομαι σε πολλά και το ε, ISDS νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο στο TTIP αυτό. Κατά την άποψή μου ούτε καν το TTIP είναι απαραίτητο, αλλά τέλο πάντων το ISDS είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και χαίρομαι που έχετε μια τόσο θαραλέα θέση. Συμφωνώ και γι' αυτό που λέτε ότι η πολυπλευρικότητα των εμπορικών συμφωνιών είναι προτιμητέα και συμφωνώ επίση, όπω προτείνετε και εσεί, να μην περιληφθεί η εκπαίδευση, η υγεία και άλλοι τομεί στο TTIP. Νομίζω ότι αυτοί οι τομεί θα πρέπει να θίγονται και θα πρέπει να συστούμε στον ελληνικό κατάλογο. Και χαίρομαι επίση που θέσατε το θέμα του αντικτύπου. Πρέπει όμω να διευκρινίσω ότι για τι αξιολογήσει ε, του τότε από την Κομισιόν έχουμε μόνο ευχολόγια και θετικέ εκτιμήσει εμείς ξέρουμε ότι αντίθετα θα οδηγήσει στην κατάρρευση του εσωτερικού κοινωνικού εμπορίου και σε αύξηση της ανεργίας. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πληγούν ιδιαίτερα από τη δικασία αυτή νομίζω ότι όλοι υπερεκτιμούμε τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει το TTIP. Γιατί στην πράξη πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χάσουν μερίδιο αγοράς εις βάρος μάλλον προ όφελο των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι για τι μικρομεσαίε είναι δικό μα καθήκον να απαιτήσουμε ένα κεφάλαιο για αυτέ που να μην περιορίζεται σε ανταλλαγή βαλτιστών πρακτικών και σε ευχολόγια. Να επιθυμίσω σε αυτού που λένε ότι το TTIP θα είναι ιδιαίτερα θετικό για τι μικρομεσαίες ότι στην πράξη μια μικρομεσαία καταρχά θα πρέπει να συμφωνήσουμε τον ορισμό οι μικρομεσαίε αυτέ είναι επιχειρήσει. Ε, με εκατομμύρια ευρώ τζίρο, 200 ας πούμε, εργαζόμενους, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ πιο μικρές. Όποιος λοιπόν ήδη εμπορεύεται με τις ΗΠΑ θα ωφεληθεί. Και εγώ θυμάμαι ότι για να ανοίξει μια αγορά δεν αρκεί να θέλουμε να το κάνουμε. Χρειάζονται επενδύσει, δομέ και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε έτσι να εφεύρουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν κίνητρα στι μικρομεσαίε. Όχι μόνο μέσω ενό αποκλειστικού κεφαλαίου βελτίστων πρακτικών. Για το ρυθμιστικό τμήμα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να υποχωρήσει χωρί δημοκρατικέ διαδικασίε από αυτή τη συμφωνία, εάν και εφόσον εγκριθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά, εκ μέρου όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών, την εμπλοκή των stakeholders, κοινωνία των πολιτών και των πολιτών κυρίω όσον αφορά τα ρυθμιστικά. Καμιά συμφωνία δεν μπορεί να συναφθεί, έστω και αν μόνο θεωρητικά θα μπορούσε να θίξει τις προγραφές ε, που έχουμε στην Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν καλά το TTIP και ότι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να το εξηγήσουμε. Εγώ λοιπόν αυτό κάνω εξωκοινοβουλευτικά, αλλά οι πληροφορίε μας θα πρέπει να είναι ισόρροπες και να μιλάνε και για τα καλά καλά και για τα άσχημα. Και όπως λέμε και στα τελικά, αν το γνωρίζεις το TTIP, μάλλον θα το αποφύγεις. Σας ευχαριστώ πάντως, θαυμάσια η έκθεση, με κάποιες πτυχές που θα μπορούσαν να βελτιωθούν και θα συμβάλλω και εγώ σε αυτό το τροπολογίες. Ευχαριστώ. So, liebe Kollegen, Kollegen, jetzt haben wir die eine Stunde. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξαντλήθηκε η πρώτη ώρα. Με τις συνομιλίες δεν έχουμε τη δυνατότητα τώρα να ακούσουμε αμέσως, αμέσως να ακούσουμε άλλους συναδέλφους γι' αυτό προτείνω στην προσεχή συνεδρίαση να συνεχίσουμε Έχουμε 12 συναδελφούς που έχουν στήσει το λόγο. 18 Μαρτίου λοιπόν και πριν να εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα έχουμε την ευκαιρία να συστήσουμε διεξοδικά τη συνέχεια. Μα πρόεδρε θέλω απλώς διαδικαστικά να θέσω το εξή και ζητώ το λόγο για ένα λεπτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Επιτροπή μας. Θέματα τόσο σημαντικά που ενδιαφέρουν όλους τους βουλευτές δίνεται το λόγο μόνο στους συντονιστές μας. Λοιπόν, τρέφω κάθε σεβασμό και εκτίμηση για τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Συχνά μας λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τους υποστηρίζω πλήρως. Αλλά, επί της ουσίας, καμία ευρωπαϊκή συνθήκη δεν ορίζει ότι στα σημαντικά θέματα το λόγο θα λαμβάνουν μόνο συντονιστές. Στο το υπενθυμίζω κύριε Πρόεδρε και το λέω γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κανονίστε και οργανώστε τη δουλειά μας έτσι, από εδώ και μπρο, ώστε οι βουλευτές να μπορούν στο σύνολό τους να εκφράζονται. Έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όλοι οι ευρωβουλευτές και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Μ' ακούτε, μ' ακούτε, μ' ακούτε. Λοιπόν, δεν μίλησαν συντονιστέ για να διευκρινίσουμε. Σκιώδη ηγητέ Γι' αυτό είχαν περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την επεξεργασία του θέματος. Τουλάχιστον μία ώρα ακόμα θα προβλέψουμε στην επόμενη συνεδρίαση και για τους βουλευτές για να συνεχίσουμε την περαιτέρω συζήτηση ώστε να έχουμε το χρόνο να τα δούμε όλα αυτά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για τις 26 Μαρτίου. Τώρα δυστυχώς όπως είπα πρέπει να διακόψω για να μεταβώ στην ακρόαση για την Ήτρε, με την Ήτρε και θα αναλάβει ο συνάδελφος με διευθύνη τις, ναι, ε, τις εργασίες μας. dear colleagues and uh, dear members and dear guests. Συνάδελφοι, φίλοι, προσκεκλημένοι. Συνάδελφοι, και προσκεκλημένοι, παρακαλώ όσοι τελειώσατε εδώ με την αίθουσα αφήστε τους υπολοίπους που έχουν δουλειά ακόμα να παρακολουθήσουν. 15. Σήμερα 15 στην ημερήσια. Έκτακτα εμπορικά μέτρα για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη δικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναστολή της εφαρμογής τους όσον αφορά τη Βοσνία Ζεβοβίνη. τον Μπετίνη ο συγητής. για τα δικά Βαλκάνια. Προτιμήσεις παράταση μέχρι το 2020. Η Κομισιόν προτείνει να αρθεί η παράταση το 16 για τη Βοσνία Ζεγοβίνη επειδή η χώρα δεν συμφωνεί για τη δικασία σταθεροποίησης και σύνεσης. Δεν λαμβάνει υπόψη της την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Να καλωσορίσω τον Εγκουαρδαβίτοβιτς, την αυτού εξοχότητα πρέσβη της Βοσνίας Ζεγοβίνης πριν συζητήσουμε το κείμενο του κυρίου Μπετίνη, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταβίδο να μα παρουσιάσει τη θέση τη χώρα του. Εξοχότα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπετίνη και μέλη τη Επιτροπή. σα ευχαριστώ να πω καταρχά και να υπογραμμίσω τη διάθεση τη Βοσνία Ερζεγοβίνης να διαπραγματευτεί την προσαρμογή του πρωτοκόλου για την ε, Συμφωνία σύνδεση. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Έχουμε μία εντολή στην αντιπροσωπεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης η οποία δόθηκε από τις ε, κρατικέ αρχές και από τον Νοέμβρη του 12 μέχρι τον Ιούλιο του 2013 η αντιπροσωπεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης συμμετείχε σε τρει γύρου διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση του πρωτοκόλου SAA. Δυστυχώς, οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να πετύχουν συμφωνία. Κατά συνέπεια, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έναρξη διαβουλεύσεων για α, ρύθμιση για επιδιαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 49 της ενδιάμεσης συμφωνίας. Το Δεκέμβριο έγινε το 13 χωρίς αποτελέσματα. Επίσης, για την φύση της συνάντησης διαφώνησαν τα δύο μέρη. Η Βοστίνα Ζεγοβίνη είναι διατεθειμένη να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ε, δραστηριότητε για την προσαρμογή της ΕΜΕΣ Συμφωνία. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιλάβει το παραδοσιακό εμπόριο στις ε, διαδικασίες ώστε να απελευθεί στις τεχνικές προσαρμογές. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια σημαντική τροποποίηση του καθεστώτος εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Βοσνίας Ερσεγοβίνης και θα μπορούσε ε, δεν θα μπορούσε μάλλον να θεωρηθεί καθαρά τεχνική προσαρμογή. Θεωρούμε ότι οι συζητήσεις πέραν των τεχνικών προσαρμογών σημαίνει ότι δεν υπάρχει τήρηση της προηγούμενη συμφωνίας. Και το SAA που υπό, υπέγραψαν 27 χώρες μέλη δεν προβλέπουν υποχρεώσει για την διατήρηση των εμπορικών ροών σε περίπτωση διεύρυνση. Από την άλλη μεριά, η Βοσνία Ζεγοβίνη από την αρχή προώθησε ένα καθεστώ ελεύθερου εμπορίου και άνοιξε τα προϊόντα τη για τα προϊόντα τη Ένωση. Η φιλελευθερωποίηση καλύπτει γύρω στι 250 γραμμέ δασμών και πάρα πολλά προϊόντα. Αλλακτοκομικά, με ζάχαρη και πολλά άλλα. Έχουμε το 3% όλων των γραμμών δασμών που καλύπτονται από αυτές τις συμφωνίες. γραμμέ οι οποίε είναι σημαντικέ για την Βοσνία Ζεγοβίνη και είναι σημαντικέ για την άπτυξη τη οικονομίας της. Η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Βοσνία Ζεγοβίνη και ΕΕ επιτεύχθηκε για να διατηρηθεί ένα πλήρε καθεστώ δασμών για αυτές τις γραμμέ προϊόντων. Ο βραδικός τομέας περιέχει ένα σημαντικό κοινωνικό στοιχείο και η παραμικρή διατάραξη του μπορεί να δημιουργήσει πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το άνοιγμα της αγοράς μας στις 28 χώρες της Ένωσης σημαίνει καταστρέφοντας τον γεωρικό μας τομέα ε, σημαίνει ότι θα έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας 3.000 ατόμων. Ε, περαιτέρω, η φιλευθεροποίηση αυτής της αγοράς σημαίνει ότι για τα προϊόντα αυτά θα Η αλλαγή στα προϊόντα αυτά θα οδηγήσουν στην υποβάθμιση της οικονομίας μας. Πάντως, η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις τεχνικές προσαρμογές της ενδιάμεσης συμφωνίας και του SAA. Όπως αναφέραμε, προτείνει η αντιπροσωπεία μας ποσοστώσεις για ψάρια, ίνο και ζάχαρη με αντίστοιχε ποσότητε εξαγών από Βοσνία Ερσεγοβίνη σε Κροατία και αντίστροφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα δεν μα έδωσε την ομοδότησή τη για αυτή την πρόταση. Λυπούμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλο που συνεχίζονται διαπραγματεύσει, υπέβαλε μία πρόταση για το 2014 αποβλέποντα το να εξαιρεθεί η Βοσνία από τον οικονομισμό που αφορά την ισχύ των ATM από την 1η Γενάρη 2015. Αυτό έχει σημαντικέ επιπτώσει σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα λόγω των θεομηνιών που είχαμε. Από την άλλη μεριά, η πρωτοβουλία αυτή τη Κομισιόν, σύμφωνα με τις ε, εκτιμήσει μα οδηγήσει σε έλλειμμα εμπορικό γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. θα πρέπει να έχουμε την ίδια μεταχείριση όπω άλλες συμφωνίε που αφορούσαν άλλες χώρε όπω την Κροατία χωρί προτιμησιακά καθεστώτα Όπω επίση, οι συμφωνίε ε, που υπάρχουν με την Σερβία. Από την προοπτική λοιπόν σκοπιά αυτή είναι σημαντικό οι δύο πλευρέ να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσει, τη δικασία διαπραγματεύσεων ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το καλό όλων μα. Κάνουμε έκκληση και ελπίζουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατανοήσουν την κατάσταση και να δώσουν οδηγίε στην Κομισιόν να συνεχίσει τι διαπραγματικέ διαδικασίε ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για όλου μα. Ενώ ε, λέγοντα μα, Ένωση, Βοσνία Ζεγοβίνη ή Βοσνία Ζεγοβίνη και Κροατία. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την πρόσφατη πρωτοβουλία τη Ένωση, η οποία επικεντρώθηκε στι ε, κοινωνικέ μεταρρυθμίσει που υποπολέμους να ενισχύσουν την οικονομία τη Βοσνία της όπω ήδη γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο τη Βοσνία της χθε υιοθέτησε αυτή τη νέα πρωτοβουλία και όλη η χώρα έχει αφοσιωθεί στο να τηρήσει και να τιμήσει τη συμφωνία τη με την ε, Ευρώπη και ίδιος ο Επίτροπος Χάν ε, καλωσόρισε αυτή την εξέλιξη. Εγώ ίδιος ε, προσωπικά Ήμουνα στην κυριολεκτική ε, Συνόδοση της Βονίας της όπου η κυρία Μογκερίνη χαιρέτησε ακριβώς αυτή τη νέα προσέγγιση, δηλαδή την οικονομική επανοικοδόμηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ως ένα είδος νέα ατζέντα για την επιτάχυνση, όχι μόνο το μπλοκάρισμα της ε, διαδικασία ομπαρική ολοκλήρωση. Σας παρακαλώ να λάβετε γνώση στο γεγονό ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταστροφή της οικονομίας μα, αλλά θα πρέπει αντίθετα να βρεθούν αμοιβαίε λύσει που θα λαμβάνουν υπόψη του τα συμφέροντα και τι απόψει και των δύο πλευρών. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι η Βοσνία Ερσεγοβίνη είναι έτοιμη να μεγιστοποιήσει τι προσπάθειέ τη ώστε να βρεθούν έγκαιρε λύσει όχι μόνο για το δικό τη συμφέρον αλλά και το συμφέρον ολόκληρη τη διαδικασία αυτή. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι είμαι διπλωμάτη λόγω επαγγελμάτος αλλά πρέπει να πω ότι θα πρέπει να προσδοκούμε στις διαπραγματεύσεις, στον επόμενο γύρο τους και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα βρεθεί μια επικοδομητική λύση ώστε να μην έχουμε διαδικασίες ε, διατησίας κάθε άλλο να επιταχύνουμε αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας Πρόεδρε και είμαι έτοιμος και στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε τη θέση της κυβέρνησής σας. Δίνω το λόγο τώρα στον εισηγητή. Θα τον πετύνει. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, έχετε το λόγο. Συνάδελφε Πρόεδρε, η έκθεση που συζητάμε πρακτικά έχει περιορισμένη σημασία εκτός για Κροατία και Βοσνία Σεγοβίνη πολιτική σημασία και επειδή αναφέρεται στους κανόνες στις σχέσεις μεταξύ χωρών της Ένωσης, της Ένωσης άλλων χωρών που βαδίζουν, που οδεύουν προς την Ένωση ή επειδή αφορά τη Βοσνία, μια χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη με υψηλή συμβολική σημασία. Για αυτούς τους λόγους στην σύνταξη της ε, γνωμοδότησης προσπάθησα να αναζητήσω συνενέσεις που αυτή τη στιγμή νομίζω μπορούν να βρεθούν. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για την γνωμοδότηση με σημαντικές συμβολές. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Λάγκ, τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, τον εισηγητή Άφετ, τον Σκιώδη από το ΕΛΚ, ΣΤΙΕ, ΕΕ, και τους άλλους κοιόδης από τις διάφορες άλλε πολιτικές ομάδες. Λοιπόν, ποιε γενικέ γραμμέ ακολουθήσαμε για, το... για την ισορροπία αυτή, η δυναμική θα τη χαρακτηρίζα, ώστε η Βοσνία να συμμορφωθεί με τους κανόνες που έχουν αποδεχτεί όλες οι υπόλοιπε χώρες των Βαλκανίων όσον αφορά την προσαρμογή στους εμπορικούς κανόνες της Ένωσης και ταυτόχρονα όμως να υπάρχει μια σημαντική όθηση της προοπτική προοπτικής προσχώρησης της Βοσνίας στην Ένωση. Η Βοσνία πράγματι δεν θα πρέπει να παραμείνει αδρανής πέντε χρόνια για να κάνει σημαντικά βήματα προ την Ευρώπη όπω κατανοήσαν κάποιοι μετά από την ανακοίνωση του Γιούγκ να μην προχωρήσουμε σε επόμενη διεύρυνση. Αντίθετα θα πρέπει να αποφεληθούμε άμεσα την τωρινή θητεία ώστε το χύτερο δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασία για την προσχώρησή της. Α πάμε τώρα στην ουσία. Η πρόταση της Κομισιόν, τροποποιώντας τον κανονισμό του 2009 τον 2015 για τα εμπορικά μέτρα τα έκτακτα, προτείνει τρία θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν μπορούν να συζητηθούν ούτε και βέβαια να αποτελέσουν αντικείμενο διαφωνίας. Δηλαδή, διεύρυνση μέχρι το 2020 του καθεστώτο του πρωτομησιακού για τι Ευρωπαϊκέ Χώρε όπω καθορίζει ο κανονισμό του 2009 αυτό επιβεβαιώνει και τη δικιά μας την πολιτική υποστήριξη και προώθηση για τη σταθεροποίηση όλης της περιοχής των Βαλκανίων. Κατά δεύτερο λόγο τη δυνατότητα διακοπής αυτών των προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων τη στιγμή όπου οι χώρες που απολαμβάνουν αυτών των σχέσεων παρουσιάζουν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ρήτρα ανθρωπίνων λοιπόν δικαιωμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ένωση επειδή αφορά τις αρχές που αφορούν την ακαιρεότητα των ατόμων και την ελευθερία τους. Και κατά τρίτο λόγο, η αύξηση της ποσότητας για, την, για τις εξαγωγές ίνων. Αντίστοιχη η ποσότητα συμμαθέως των υπόλοιπων χωρών Βαλκονίων. Εδώ η Κομισιόν αντιμετώπισε άλλο ένα λεπτό ζήτημα ότι μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από την προσχώρηση σε αυτήν η Κροατία η Βοσνία δεν αποδέχτηκε την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων στα πλαίσια της ενδιάμεση συμφωνία ώστε να υπάρχουν παραδοσιακέ προτιμησιακέ ε, συναλλαγέ μεταξύ Κροατία και Βοσνία. Όπω καθορίζει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών ΣΕΦΤΑ. Στην περίπτωση όπου η Ένωση και η Βοσνία δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν όσον αφορά τι εμπορικέ παραχωρήσει, συμφωνία που εμεί ε, επιθυμούμε, οι προτιμήσει που θα δοθούν στην ε, Βοσνία χάρη στο 2015-2009 θα αρθούν από την 1η του Γενάρη 2016. Εάν στη συνέχεια η συμφωνία επιτευχθεί, οι προτιμήσεις αυτές θα επαναφερθούν. Όπως βλέπετε, πρόκειται μια ήπια πίεση, επειδή ακριβώς η αξία αυτών των προτιμήσεων ε, των εμπορικών αξιολογείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίω Εξάλλου, Η άρνηση προσαρμογή της Βοσνίας οδηγεί στο ότι τα κροατικά προϊόντα τα οποία έχουν προτίμηση του βοσνιακού πληθυσμού να κοστίζουν στον πληθυσμό της Βοσνίας πολύ περισσότερο λόγω των δασμών στους ε, οποίους υπόκειται η ίδια η Βοσνία μετά από την προσχώρηση της Κροατίας. Η Βοσνία λοιπόν δεν αναγνωρίζει την νομιμότητα αυτών των ετοιμάτων και λέει ότι υπάρχει ισχυρό πλήγμα για την οικονομία της σε περίπτωση που τα αποδεχτεί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά σαφής ε, αρκετά σαφή τα επιχειρήματα της Κομισιόν. Η προσαρμογή που στήθηκε από τη Βοσνία ήδη έγινε αποδεκτή από τις υπόλοιπε χώρες της περιοχής κατά τη διάρκεια της, προσαρμογής, της, προσ, της προσέγγισης τους προς την Ευρώπη. Κωσυφοπέδιο, Αλβανία κτλ. Και είναι κάτι το οποίο διέπει τι συνήθειε διαδικασίε διεύρυνση τη Ένωση. Δεύτερο, υπάρχει μια λογική κατεπίγουσα. Δηλαδή, αν εξάγουμε απελευθερωμένα προϊόντα στην Βοσνία, α πούμε 100 και με 27 χώρε, από τη στιγμή όπου προστίθεται μια άλλη χώρα, όπω η Κροατία σε αυτή την περίπτωση, οπότε πάμε από τα 27 στα 28 μέλη, αν λοιπόν το μέτρο το, του 100 παραμένει το ίδιο και δεν προσαρμόζεται, τότε αυτό προποθέτει μία ζημιά για τον τελευταίο αφιχθέντα και όλη την Ένωση. Και αυτό ακριβώ θεωρεί η Κομισιόν ότι η απαραίτητη προσαρμογή στην ουσία αποτελεί ένα copy-paste του όγκου και της τυπολογίας των συναλλαγών με την υποσμία που λαμβάνουν χώρα μετά τη διεύρυνση σε 28. Θα πρέπει δηλαδή απλά και μόνο να αναγνωριστεί στα πλαίσια συνέμεσης συμφωνία μεταξύ Βοσνία και Ένωση και αυτό το οποίο ανταλλασσόταν στα πλαίσια του παραδοσιακού εμπορίου μεταξύ Βοσνίας και Κροατίας. Δηλαδή, μεταξύ Βοσνίας ε, και Ένωσης των 27, εάν ας πούμε συμβολικά και πάλι είχαμε ανταλλαγή 100, εάν μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας συναλλασσόταν 10, με την είσοδο τη Κροατία που αυξάνει τις 28, δεν μπορεί να παραμείνει 100 αυτό το μέτρο, θα πρέπει να προσθέσουμε το 10 και να πάμε στο 110. Διαφορετικά βεβαίως υπάρχει αλλίωση των ισορροπιών. Τέλος, και απελευθέρωση κάποιων προϊόντων που αυτή τη στιγμή προστατεύονται από την υποσυνία στις ε, συναλλαγές με την Ένωση θα γίνει για τις ποσότητες που ήδη προβλέπεται για τι παρουσιακέ συναλλαγέ μεταξύ και Βοσνίας πριν από την προσχώρηση Κροατία στην Ένωση. Καταλήγοντα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα από την Βοσνία, πέραν δηλαδή από τι συνθήκε που προπήρχαν τη εισόδου τη Κροατία στην Ένωση. Φαίνεται λοιπόν λογικό και θεμητό αυτό που έκανε η Κομισιόν για την άρση ως μέσο ήπιας πίεσης για την επίτευξη λογικής συμφωνίας. Ας πέσουμε τώρα στο δεύτερο σημείο που ανέφερα προηγουμένως, το πολιτικό ζήτημα. Ο μηχανισμός που προτείνεται σήμερα περισσότερο από όσο ποτέ πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος όθησης προς δέσμευση παρά ως απειλή για κυρώσεις. Σήμερα είχαμε εξελίξεις όσον αφορά την ε, προοπτική προσχώρηση της Βοσνίας Ζεγοβίνης στην Ένωση. Αναφέρθηκε ο πρέσβης προηγουμένως αυτά και τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Ξέρουμε ότι η Βοσνία αντιμετωπίζει δυσκολίες ε, με τις μεταρρυθμίσεις. Μαστίζεται από διαφθορά και από διοικητική αταξία. Παρουσιάζει ε, δομές περίπλοκες και έχει υποστεί βεβαίως και θεομηνίες αλλά και άλλες ιστορικές ιστορικά δεινά. Ξέρουμε όμως ότι μπορεί να τα καταφέρει η Βοσνία, ο λαός της προσβλέπει με ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διατεθειμένος να καλλιεργήσει την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει μόνα της, μόνη της, αν την εγκαταλείψουμε στην τύχη της ε, και σε επικίνδυνες εξωτερικές επιρροές. Εδώ υπάρχει μια προφανής δική μας ευθύνη. Αν θέλουμε και για μας και για την Ευρώπη να αποφύγουμε άλλες περιπέτειες. Γι' αυτό ακριβώς κρίνω μεγάλη σημασία στη νέα προσέγγιση που η Κομισιόν και το Συμβούλιο επέλεξαν για τις σχέσεις με την Βοσνία, κυρίως μετά από την ε, πρωτοβουλία της κυρίας Μογκερίνη. Δηλαδή να αντιστρέψουμε την πυραμίδα, να μην ζητήσουμε αμέσως από την Βοσνία να αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα ζητήματα με τα αποτελέσματα τα πολύ έτσι ε, ισχνά όπως ξέρετε και αντίθετα να ζητήσουμε να κάνουν πρακτικά, εφικτά και απτά βήματα. Αυτή η προσέγγιση που συζητήθηκε στο Σεράγεβο σε μέγιστο πολιτικό βοσνιακό επίπεδο το Δεκέμβριο 2014 ήδη είχε ένα αποτέλεσμα θετικό. Ένα έγγραφο δηλαδή ξεκάθαρων δεσμεύσεων επίσημων που προσυπόγραψαν οι ηγέτες, οι κυριότεροι ηγέτες της χώρας ώστε να υλοποιηθούν χωρίς, δισταγμή, χωρίς δισταγμούς τα απαραίτητα βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρώντας τις αρχές και τις αξίες οι οποίες αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έγγραφο υιοθετήθηκε επίσημα χθες με την παρουσία της κυρίας Μοκερίνη από τις δύο πλευρές του Βοσνιακού Κοινοβουλίου. Ε. Αυτό επιτρέπει την θέση σε εφαρμογή οριστικά της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης και Σταθεροποίησης της Βοσνίας ε, με την Ένωση σημαντικό βήμα προς την προσχώρηση. Σήμερα για τα, για τα εμπορικά ζητήματα λοιπόν δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το πλαίσιο εξελίξει και το χαρακτηρίζω ως όθηση, ως κίνητρο αυτή την έκθεσή μας, ώστε απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις να βοηθήσουμε την Βοσνία να πετύχει το πιο στρατηγικό και πιο σημαντικό στόχο για αυτήν, δηλαδή την προσχώρηση στην Ένωση. Για τη σημασία λοιπόν που παρουσιάζουν αυτά τα πολιτικά στοιχεία, προς, αποφάσισα να προσθέσω στην έκθεσή μου ένα, ένα εκτιμώντα 7. Δηλαδή ζητώντας την επίλυση της διαμάχης με τη Βοσνία με αμοιβαία αποδεκτή λύση. Θεώρησα ότι είναι σημαντικό να προσθέσω το διατακτικό μία σαφή έκκληση στην δέσμευση της Ένωσης για την προοπτική προσχώρηση της Βοσνίας, όπως ακριβώς καθορίζουν τα συμπεράσματα του, Υπουργείου, του Συμβουλίου Εξωτερικών του, της, 5ης Δεκέμβρη 2014. Και θα ήθελα να εθετήσω επίσης και την ε, πρόταση του συναδέλφου Πρέντα να κάνουμε θετική τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνοντα την πιο υποχρεωτική, πιο δεσμευτική. Τέλο, προτείνω να εφαρμόσουμε την διαδικασία με κατεξουσότηση πράξη για την άρση των προτιμήσεων, αν δεν τελειθούν οι, οι προποθέσει που θέτει η Ένωση στι εμπορικέ συμφωνίε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους της Κομισιόν για να αξιολογηθεί το κατά πόσο οι προτιμήσεις αυτές έχουν τηρηθεί. Οπότε θα πρέπει να έχουμε αξιολογήσεις που πηγαίνουν πέρα της απλής εφαρμογής, οι οποίε όμως είναι υποκειμενικές, επειδή ακριβώς το πεδίο της ε, άρσης δεν έχει προσδιοριστεί. Οπότε, δηλαδή, η Κομισιόν μπορεί να κάνει άρση αυτών των προτιμήσεων μερικώς ή γενικώς. Είναι απαραίτητο πάντως να εμπλακούν και οι σύνομοθέτε και να υπάρχει μια σωστή επιτήρησή του. Θεώρησα να... ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε και τι εκτελεστικέ πράξει, τι υπόλοιπε διατάξει του βασικού κανονισμού που έχουν πιο περιορισμένο εύρο και τα κριτήρια συμμόρφωση. Εκεί τα κριτήρια είναι πιο αντικειμενικά. Αυτό που ανέφερε ο κ. Πρέντα από την ΑΦΕΤ νομίζω ότι εκφράζει μια ισορροπία σε σχέση με ε, άλλα ζητήματα όπως εργασιακά δικαιώματα, περιβάλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διατύπωση της Κομισιόν, αλλά παρόλα αυτά είναι ανοιχτός για συζήτηση με τους ε, συναδέλφους μετά από αυτά που έχουμε και στην ΑΦΕΤ. Από σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η διαδικασία της έκθεσης αυτής σύμφωνα με μια διαβάθμιση την οποία θα σας κοινοποιήσω διανέμοντα την έκθεσή μου που παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα βήματα μέχρι την κατάληξη στην Ολομέλεια, στην δεύτερη Ολομέλεια του Απρίλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την συνεργασία και θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στο ευαίσθητο τη συζήτησή μας από όπου θα πρέπει να ανακύψει μια σοβαρότητα στις πράξεις μας και στην δυνατότητα που θα έχει η Ευρώπη να αξιοποιεί την πολιτική προστεθέμενη αξία η οποία είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις που έχουν μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and... Uh, πολύ σας ευχαριστούμε και τώρα να ακούσουμε τους κοιόδες ε, εισηγητές από το ΕΛΚΟ κύριο Στία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον πρέσβη από την Βοσνία Ζεγοβίνη καθώς και τα μέλη της αποστολής. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το συγκερασμό των απόψεων που κατάφερε ε, καταλήγοντας ένα ε, ισόρροπο κείμενο. Ευχαριστούμε. Από πλευρά ΣΕΛΚ Υποστηρίζουμε την επέκταση των πρωτεμισιακών διατάξεων σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, φαίνεται να είναι η ορθότερη προσέγγιση αρρωγή προς αυτές τις χώρες, ώστε να προετοιμαστούν αυτές οι χώρες και να ακολουθήσουν το οδό της ε, προσχώρησης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως προς τις τροπολογίες του εισηγητή, όταν ε, μιλάμε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις παραβιάσεις ε, και μιλάτε για κατεξουσιοδότηση πράξη, πιστεύω ότι είναι σημαντικό το μέτρο και θέλουμε να το υποστηρίξουμε. Επίσης, συμφωνούμε με τον εισηγητή πως για τη Βοσνία Ζεγοβίνη θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενθάρρυνση αυτό το μέτρο. Προσβλέπουμε στην ε, σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις αρχές της ε, ε, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγγνώμη, πριν λήξει το 2015. θέλουμε να τεθεί σε ισχύ πριν το 2016 για την επέκταση των προτιμησιακών καθεστώτων είναι σημαντικό να τροποποιηθεί και η διάμεση συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Κροατίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όπως έγινε και από όλες τις υπόλοιπες ε, γειτονικές χώρες και από την Κροατία ε, πριν την προσχώρηση σε σχέση με την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Και τουλεχθέντως θα υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση του εισηγητή σε σχέση με την προσθήκη αιτιολογικών σκέψεων ε, που ξεκάθαρα διευκρινίζουν πως υπάρχει σαφής πολιτική υποστήριξη για να ακολουθήσει η Βοσνία Ζεγοβίνη την οδό τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Έχετε τη δήλωση τη κυρία Μουγγερίνη, αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι οι δηλώσει των αρχών τη Προεδρίας και τη κοινοβουλευτική συνέλευση της Βοσνίας Ερσεγοβίνη. Όπως είπε και ο Πρέσβη, είναι πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αυτά τα βήματα που γίνονται τώρα. Αναμένουμε το επόμενο βήμα με την τροποποίηση της ενδιάμεσης συμφωνίας επιπροσθέτως. Ως τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε, κυρίως θα φέρουμε επί της μορφής κάποιων τροπολογιών και όχι επί της ουσίας. Μία αιτιολογική σχέση που πρότεινε ο εισηγητής παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να, συντομε... να συντμηθεί Η διατύπωση να μην ε, συνδέεται με συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου διότι πιστεύουμε ότι ε, πιο μακροπρόθεσμα θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση στη Βοσνία Ζεγοβίνη και θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη διατύπωση τόσο ώστε να γίνει πιο διαχρονική. Είναι τυπικά όμως, όπως είπα, αυτά τα ζητήματα, όχι ουσιαστικά. Ε, υποστηρίζουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το κείμενο που μας ε, υπέβαλε ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το κατάλογο των σκιωδών έχουμε τον Paul Looms δεν τον βλέπω όμως, τον Όλι Ρεν. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Εγώ θα σας διαβάσω την έκθεση του εισηγητή από πλευράς ε, του ECR. Λέει εδώ ότι ελπίζουμε πως οι σε αρχές της Βοσνίας της Ζεγοβίνης θα δράξουν την ευκαιρία για να υιοθετήσουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για την σταθεροποίηση, τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και την ενδιάμεση συμφωνία στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και υπέρ των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων. Για την τροπολογία τώρα, σε σχέση με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα βρούμε μια συμβαστική λύση σε σχέση με την πρόταση της ΑΦΕΤ και τέλος η τροπολογία του εισηγητή για τις πράξεις εξουσιοδότηση θα ήθελα, θα ήθελε δηλαδή ο εισηγητής να ξέρει ποια είναι η άποψη της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου εάν συνάδει αυτό με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από το σχέδιο εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σακέ. Άλτε, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ολυρέν ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ε, ζητά συγγνώμη. Κάποια λόγια να πω και εγώ από πλευρά του. Για τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα πιο συγκεκριμένα προτείνει να διατηρηθεί η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις. Σε περίπτωση παραβιάσεων αυτό είναι ευκολότερο να αποδειχθεί. Ε, αλλιώς αν έχουμε ευρύτερο ορισμό ε, θα ε, αλλάξει η κατάσταση. Ο κύριος Ολιρέν θεωρεί ότι με έναν ευρύτερο τέτοιο ορισμό θα δυσκολευτούν οι ίδιες οι αρχές της Βοσνίας της Ζακοβίνης ε, για τη δίωξη. Καλό θα ήταν να παραμείνουμε στα εσκαμμένα και να μην εφεύρουμε κάτι καινούργιο. Για την αιτιολογική σκέψη 7 θα πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση για τη διατύπωση. Εκεί λέμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν κοινώ αποδεκτέ λύσει για το διασυναριακό εμπόριο και την ενδιάμεση συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βοσνία Ζεγοβίνη, τι σημαίνει κοινώ αποδεκτέ διατάξει σε μεγαλύτερη ευελιξία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Γιατί όταν οι Αργεντινοί είπα θα ζητήσουν νέε υπολογιστικέ μεθοδολογίε σε αντίστοιχε περιπτώσει, πού σε τι θα μα οδηγούσε κάτι κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ρεν ε, αντιπροτείνει να καταθέσουμε άλλη τροπολογία να διατυπώνοντας την ετολογική σκέψη και να λέμε θα πρέπει να βρουν μία λύση μετά το διορισμό της νέας κυβέρνησης ή κάτι τέτοιο, βάση περιπτώσει. Για τη μεθολογία υπολογισμού προτείνει να χρησιμοποιήσουμε αυτή που ισχύει σε άλλες περιπτώσεις ε, μια εναλλακτική διαφορετική μεθοδολογία θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο σε σχέση με τρίτε χώρε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί σα ευχαριστούμε για την ΚΟΕ Ουδή. Πράσινη. Ο κύριος Μπίχνερ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σχολιάσω ε, ε, κάτι που αναφέρεται στην διαλογική ε, έκθεση. Λέτε εκεί πως θέλουμε να υποστηρίξουμε τον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της Βοσνίας και Σα Σας ευχαριστώ για τη διατύπωση. Ξέρετε χθε. Η Βοσνία έκανε ένα ε, πολύ σημαντικό βήμα, ο πρέσβης το ανέφερε εξάλλου αυτό, πολύ ωραίο, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Δεν επαρκούν οι διαπραγματεύσεις ε, στο σημείο που έχουν φτάσει τώρα. Δεν μπορούμε να ε, υπεραπλουστεύουμε την κατάσταση ε, είναι καταρακωμένη η οικονομία της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ε, ξέρετε ότι οι, πολιτικές, οι κοινωνικές ανταραχές ήταν ιδιαίτερα έντονες ακριβώς λόγω της ικτρής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία και δεν μπορούμε λοιπόν να εξισώσουμε τη Βοσνία με άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Σας καλώ λοιπόν κατεπηγόντας να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και να κοιτάξουμε με προσοχή τις αιτίες. Τα τρία εκατομμύρια στις πληρωμές για μένα είναι μάλλον αμφίβολης ποιότητας στοιχείο. Εάν δούμε εισαγωγέ και εξαγωγέ. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να κοιτάξουμε και αιτίε ενδεχομένω. Α μην κάνουμε λοιπόν δυστικές κινήσει. Ας δώσουμε στην υπόθεση τον χρόνο τη α διαπραγματευτούμε του όρου έντιμους και ισότιμους. Για μια λύση που θα είναι προ το καλό των πάντων. Σα ευχαριστώ. Ευρωπαίοι των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών δεν βλέπω να στον το λόγο. Άρα κλείσαμε τη σειρά των σκιωδών. Αν θέλει κανεί άλλο. Α, ο κύριος Δερικνώτη. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Μπερτίνη. Κάνει πολύ καλή δουλειά ως εισηγητής. Αναζητεί συνένεση μεταξύ των ομάδων. Εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας συμφωνώ με τις ανησυχίε του Όλη Ρεν. Πρέπει να πω, δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητούμε λύσει λύσεις ad hoc Εμένα με ενδιαφέρει να ακολουθηθεί η παραδοσιακή μέθοδος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπολογισμού. Το... του κόστος. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνουν όλες τις προσαρμογές για να βρούμε μια λύση με την Κοσμή. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια τρίτη χώρα να κάνει επιλεκτικές σχέσεις με μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ σωστά υπόθηκε ότι αν κάνουμε εξαιρέσει για μια χώρα, οποτεδήποτε μια χώρα αποφασίσει να απορρίψει την πρώτη διεύρυνση στο μέλλον, θα έχουμε πολύ σοβαρέ δυσκολίε. Είμαστε μία και μία ένωση, Το 28 κρατημέλη πρέπει ένας εξωτερικός εταίρος να τα δέχεται με τους ίδιους όρους. Βεβαίως, τούτου λεφθέντος θα πρέπει να δούμε με προσοχή την υπόθεση της Βοσνίας. Άλλοι μέλη του Κοινοβουλίου δεν βλέπουν στον το λόγο. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την ε, ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. και χαιρόμαστε φυσικά ιδιαίτερα που υποστηρίζει η έκθεση την πρότασή μας σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υποστηρίζει την πρόταση για την διεύρυνση του πρωτομησιακού καθεστώτος ε, σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ε, εκτός και να καταλήξουμε σε ε, ξεχωριστή συμφωνία για εμπορικές εκχωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ελπίζουμε. Όντως, να μπορέσει να ξεβρεθεί μια συμφωνία, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να ανασταλεί η ισχύ των προτιμησιακών καθεστώτων. Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε, έχουν γίνει τρεις ήδη διαπραγματεύσεων που απέτυχαν διότι οι βοσνιακές αρχές δεν δέχονται την αρχή ε, του παραδοσιακού εμπορίου, όπως σωστά είπε ο εισηγητής. Αυτό, αυτή η έννοια ε, είναι απλή, ε, όπως εξήγησε και ο εισηγητής. Βλέπουμε το μέσο όρο για τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με την αύξηση των ποσοστώσεων και των δύο μερών. Εξάλλου, αυτή έχει γίνει δεκτή από όλες τις χώρες των, υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και έχει γίνει δεκτό μεθοδολογία υπολογισμού από όλες τις χώρες που το προσχωρήσουν. Η κυρία Κράκο και ο κύριος Μάρτιν ε, ξέθεσαν πολύ σωστά τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να δεχτούμε κάτι διότι θα δημιουργηθεί πολύ κακό προηγούμενο για την πιθανή αναστολή των προδημησιακών καθεστώτων. Αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κύρωση, αλλά ως ε, ενθάρρυνση προς την Βοσνία, ε, ως κίνητρο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλουμε ε, τα 307 εκατομμύρια σε δασμολογικά τέλη να χαθούν για την Βοσνία, όμως θυμάστε ότι η Κροατία είχε αντίστοιχες απώλειες, μάλλον υψηλότερες απώλειες διότι μιλάμε για μείωση 20% των εξαγών προς τη Βοσνία και απώλεια 70 εκατομμύριων ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές ετησίως. Η Σλοβενία και η Αυστρία επίσης επηρεάζονται από τη μη προσαρμογή της Βοσνίας σε αυτές τις διατάξεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο πρέσβης αναφέρθηκε σε, στην αρνητική κατάσταση και στην οικονομία της χώρας. Μην ξεχνάμε όμως ότι μαζικά ε, ε, ε, ε, επικουρείται η Βοσνία Ζεγοβίνη από την Ευρωπαϊκή Βοήθεια. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει λάβει 600 εκατομμύρια από εμά και είναι ασύμετρα μικρή η πρόσβαση στην αγορά που έχει χωρίσει μέχρι στιγμή η Βοσνία. Με τον διορισμό της νέας κυβέρνησης ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα επανέλθει σε επικοδομητικές διαματεύσεις η Βοσνία, ώστε να μην χρειαστεί να αναστείλουμε την ε, ισχύ των προτιμησιακών καθεστώτων ε, που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή η Βοσνία. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεβίνιαν για να ολοκληρωθεί και αυτό το σημείο, ας στραφούμε στον συγκεκριτή μας, ο κύριο Βετίν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Στο θέμα αυτό, στο όλο αυτό το θέμα βλέπω να συμφωνούμε όλοι ως προς τις τοποθετήσεις εκθέσεως. Και προχωρώ στα ερωτηματικά που διατυπώθηκαν. Αν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω χρόνο στην Βοσνία. Μα υπάρχει ο χρόνος ακόμα. Δεν μιλούμε για άμεση άρση της συμφωνίας. Η άρση στην οποία αναφερόμαστε πρόκειται να εμφανιστεί ένα χρόνο μετά. Οπότε υπάρχει χρόνος να βρεθούν λύσεις. Η συζήτηση αυτή που κάνουμε έχει γίνει προκαταβολικά και εν ώψη των εξελίξεων και των αριθμών που έχουμε, των στοιχείων που έχουμε. Και υπογραμμίζω ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό κλίμα που επιτρέπει να φτάσουμε στο κλίμα αυτό. Γιατί δεν θα ήθελα να χάσουμε μέσα από τη συζήτηση το φεγγάρι και να κοιτάμε το δάχτυλο όπως τα λέγαμε χαρακτηριστικά. Και όπως τα λέγαν ικανότεροι από ότι εγώ ε, στην πολιτική ιστορία το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν θέλουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον και να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον με ένα κλίμα μεγαλύτερης συνένεσης και συνεργασίας μεταξύ της Βοσνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τυφλώνικο μόνο αυτό θέμα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγράφω πρόταση του συναδελφού Πρέγκαντα που μιλούσε για ένα πιο έτσι αυστηρό, δεσμευτικό χαρακτήρα αυτής της παραμέτρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα δούμε πάντως τις τροπολογίες και νομίζω ότι κάλλιστα εδώ θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε λογικούς συμβασμούς. Όταν εγώ χαρακτηρίζω ως αποδεκτό μιλώντας για λύση αποδεκτή λύση αναφέρομαι στο διάμεσο κείμενο που είναι η νομική βάση του κανονισμού μας. Και μπορώ να σας πω ότι αποδεκτό για μένα αυτό ακριβώς σημαίνει. Εντάξει, μετά θα πρέπει να παληθεύσουμε ονομασιολογικά και τεχνικά τι συμβαίνει. Αλλά αποδεκτό συμβαίνει, σημαίνει αυτό ακριβώς. Ότι δεν μπορούμε να ζητάμε τίποτα άλλο από τη Βοσνία πέραν από το άθροισμα των συναλλαγών που προϋπήρχαν δηλαδή Ένωση συν παρουσιακές συναλλαγές την εσκορατία. Αυτό ο ριζογός αποδεκτό. Αλλά βέβαια θα πρέπει να υποστηρίζεται από αριθμού, από στοιχεία, τεχνικέ αναλύσει, ουξουμούξου, που είναι αρκετά δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή. Ατύπως, ατύπως κάτι υπάρχει αλλά πρέπει να εμβαθύνουμε εδώ τεχνικά. Πάντως, αποδεκτό ως σημείο καταλεκτικό και ισορροπίας, αυτό για μένα σημαίνει. Κατ' η πράξη, η νομική υπηρεσία έδωσε μια γνωμοδότηση θετική. Επειδή μιλάμε για μια θετική γνωμοδότηση που αφορούσε αντίστοιχη περίπτωση, για τις σχέσεις μεταξύ σημερινού Ε. Οπότε νομίζω κάλλιστα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδό που επιτρέπει σε κάποια ζητήματα τόσο, τόσο ευαίσθητα να έχουμε έτσι μεγαλύτερη μπλοκή και συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ τον εισηγητή. Προθεσμία για τις προπολογίες ε, αύριο το μεσημέρι. 25 Φεβρουαρίου. Και έτσι κλείνουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και ευχαριστούμε τον πρέσβη, τον, σκιο, τον εισηγητή, του και όλους εισηγητές. Σημείο 16. Ανταλλαγή απόψεων για τι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ με τον πρέσβη του Βιετνάμ, και τον επικεφαλής της Πραγματευτικής Ομάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ επί τη βάση ψηφίσματος της Επιτροπής μας τον Απρίλιο του 2014. Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί κατά τρόπο ιδιαίτερα δραστήριες διαπραγματεύσει. Έγινε ένα πρώτο γύρο από τι 19 έω 23 Ιανουαρίου φέτο στι Βρυξέλλε. Δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων προβλέπεται το Μάρτιο στο Βιετνάμ. Μας θυμάται με την παρουσία του ο νέο διοριστή πρέσβη του Βιετνάμ, ο ξεχωριστό κύριος Wong, τον οποίο και ορίζω στη συνεδρίασή μας. Παρουσία και του επικεφαλής της πραγματευτικής ομάδας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μάουρο Πετρουτσόνε. Καλώ τον κύριο Πετρουτσόνε πρώτα, επικεφαλής της πραγματευτικής ομάδας, να παρουσιάσει τις εξελίξεις της πραγματεύσης με το Βιετνάμ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και με χαρά επιστρέφω στην Επιτροπή για να ενημερώσω τους βουλευτές σας για τις σημαντικές αυτές διαπραγματεύσεις και τις εξελίξεις τους. Με την αδειά σας, Πρόεδρε, θα είμαι όσο το δυνατόν πιο λακωνικός για να υπενθυμίσω που βρισκόμαστε στη διαδικασία και να απαντήσω σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχουν βουλευτές. Ξεκινώ λοιπόν. Υπενθυμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργό Τζον του Βιετνάμ στην ε, επίσκεψη του Βρυξέλλες πέρυσι, όπου συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μπαρόζο τότε, μας είχε διαβεβαιώσει ότι προχωρούν καλά οι σχέσεις, ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να στοχεύουν στην ολοκλήρωση των προσεχών μηνών. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργό Τζόγκ στη συζήτηση και αναμένουμε έναν ορίζοντα περί τους έξι μήνες για να δούμε εάν και πώς μπορούν να προχωρήσουν οι πραγματεύσεις. Οι εταίροι μας από το Βιετνάμ νομίζω είχαν σαφή αντίληψη του γεγονότος ότι ε, όσο το δυνατόν νωρίτερα θέλαμε, ήθελε η ευρωπαϊκή πλευρά να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Όσοι είστε όμως τις διαπραγματεύσεις για σχέση ελευθερού εμπορίου, η ουσία πάντα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ταχύτητα. Δεν βιαστήκαμε δηλαδή να συνάψουμε πάση θυσία μια τέτοια συμφωνία. Μάλιστα με χαρά μπορώ να υπογραμμίσω ότι και η βιετναμέζικη πλευρά ε, δεν αφισβήτησε ποτέ την επιλογή αυτή, υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις ώστε να είναι στο δυνατόν πιο ουσιαστική η συμφωνία. Δεν είναι ευκαιρές, βέβαια να, να εξασφαλιστεί μια φιλόδοξη συμφωνία με μια χώρα αναπτυσσόμενη με τα χαρακτηριστικά του Βιετνάμ. Πάντως οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές τις σχέσεις αυτές. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα που πρόσφατα εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έχει υψηλό επίπεδο προσήλωσης και απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών. Υψηλό πολύ για χώρα αναπτυσσόμενη. Έχει πιστεύω πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις περισσότερες από τις γειτονικέ χώρες στην Νοτιοανατολική Ασία. Έχει μακροχρόνια προσήλωση στο στόχο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και με στόχο τις εμπορικές συναλλαγές κατά τρόπο, που θα διεξάγονται κατά τρόπο συνεπή και παράλληλο με την εσωτερική μεταρρύθμιση πράγματα τα οποία για μας αποτελούν την βελτιωτική εγγύηση για επιτυχή έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε λοιπόν αισιόδοξοι ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν και να σταθούν επιτυχία σύντομα. Ως προς τη διαδικασία θα υπενθυμίσω αυτό που είπατε και εσεί, τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων τον Ιανουάριο, τον προβλεπόμενο για το Μάρτιο στο Βιετνάμ. Στη συνέχεια πρόκειται να καταγραφεί ε, σε συνεργασία με τους Βιετναμέζους που έχουν φτάσει διαπραγματεύσεις, τα επιτεύγματά τους. Και αυτό μπορώ να πω, ύστερα από τις τελευταίες μου επαφές με τον συνομιλητή μου, συνομιλητή μου από Βιετνάμ, μπορώ να πω ότι είμαστε αισιόδοξοι για μια πιο ταχεία ε, πορεία. Δεν μπορώ δυστυχώς να είμαι πιο σαφής από αυτό, αλλά ξέρετε ε, είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε διαπραγματευτεί να ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ας περάσουμε όμως τώρα στην ουσία. Δεσμολογικές διαπραγματεύσεις για τις συναλλαγές σε προϊόντα. Το, το Βιετνάμ έχει επιδείξει ψηλό επίπεδο φιλοδοξίας με την πρώτη δασμολογική προσφορά συμφώνησαν την απελευθέρωση κατά 85% των δεσμολογίων τους οι δύο πλευρές, άρα μας έχουν μείνει τα υπόλοιπα 15% και ενώ δεν είναι πιθανό να φτάσουμε σε 100% απαλλαγή από τους δασμούς ε, για όλα τα προϊόντα, θα είμαστε πολύ κοντά στο 100%, κάτι το οποίο θα αποτελεί μάλιστα και ανευπροηγουμένο εξέλιξη σε με αναπτυσσόμενη χώρα το μέγιστο που έχουμε φτάσει με την ε, Νότια Κορέα και τον Καναδά όπως ξέρετε ε, είχε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αλλά για πρώτη φορά θα έχουμε α, ισοδύναμο υπολογίζουμε ποσοστό και επίπεδο κατάργηση τασμών με χώρα αναπτυσσόμενη. Φυσικά και οι δύο πλευρέ έχουν μια σειρά από ευαίσθητα προϊόντα, αυτά θα προστατευτούν πλήρω. Έχουμε επίση συμφωνήσει ότι και για αυτά τα προϊόντα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προσφέρουμε ε, μια λογική, μια εύλογη πρόσβαση στην αγορά. Οι δεσμεύσεις GATS του Βιετνάμ είναι υψηλής ποιότητας. Η συζήτηση συνεχίζεται εκεί που είχε σταματήσει πριν από 10 χρόνια όταν σταματήσαμε τις ε, διμερείς διαπραγματεύσεις της αγοράς ενώπιστον ε, της προσχώρησης στον ΠΟΕ και μπορούμε να συνεχίσουμε για το διμερές επίπεδο. Δεδομένης της ε, δέσμευσης στην ΚΑΤΣ του Βιετνάμ είναι πολλοί οι τομείς πιστεύουμε όπου μπορούμε να δούμε την αλλαγή γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς ε, στην οικονομία του Βιετνάμ που δεν έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες μιας ε, σύμβασης ελεύθερων συναλλαγών στην πραγματεύση της ΚΑΤ. Στις διαπραγματεύσεις δεν με μια αναπτυσσόμενη χώρα είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε όλα τα ζητήματα γιατί πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη και η πιο ευάλωτη θέση του εταίρου μας γιατί δεν θα πρέπει να επιδεινώνεται ε, ή να πιέζεται η θέση του εταίρου αναπτυσσόμενου κράτους στο να βελτιώσει την διαπραγματευτική του θέση. Αλλά από την άλλη θέλουμε να έχουμε και καλές συνθήκες συναλλαγών με του εταίρους μας και νομίζω ότι αυτό είναι το πράγμα με το οποίο και το Βιετνάμ προσεγγίζει τι διαπραγματεύσεις. Επενδύσεις κυρίως στο τομέα εκτός των υπηρεσιών. Επίσης έχει δηλώσει βούληση για ε, ταχεία πρόοδο και κάλυψη του χαμένου εδάφου σε σχέση με την απελευθέρωση των υπηρεσιών το Βιετνάμ σε σχέση με το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπως τις περιγράφουμε στις διμερείς σχέσεις. Η Δημόσια Συμβάση είναι ένα πολύ σημαντικό, όπως ξέρετε, θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα ταχύτατα αναπτυσσόμενη το Βιετνάμ με ανάγκες μεγάλες σε υποδομές και ανάπτυξη ε, τομείς που, όπου εν γέννη οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι πολύ ανταγωνιστικές ωστόσο δεν έχει τέτοιο, τέτοια εμπειρία και ιστορικό διαπραγματεύσεων διεθνών στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων το Βιετνάμ και άρα αυτό το κόμμα των διαπραγματεύσεων είναι πολύ περίπλοκο ταυτόχρονα επαναλαμβάνω ότι σημειώνουμε και πάλι την πολύ σημαντική προσήλωση του Βιετνάμ. Γιατί οι εταίροι μας αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο μπορούν να βελτιώσουν το εσωτερικό, το εθνικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις με, με τα ωφέλη που γνωρίζουμε για καλύτερες συμβάσεις προς όφελος των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών, ε, διαφάνεια και απρόσκοπτη εκτέλεση των συμβάσεων. Εν γέννη, το θεματολόγιο μας είναι αντίστοιχα ε, διατυπωμένο όπως έχουμε και με τις άλλες χώρες, δηλαδή καλύτερη συνεργασία, διαφάνεια. Ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ αναφέρονται και στις κρατικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι από την αρχή των διαπραγματεύσεων μπορέσαμε να προσδορίσουμε μια βασική φιλοσοφία και να συμφωνήσουμε σε αυτά που ορίζει άλλωστε και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δηλαδή δεν παρεμβαίνουμε σε θέματα κυριότητας, ιδιοκτησίας δηλαδή του κράτους για τις επιχειρήσεις. Διαφυλάτουμε το, την αρχή της ουδετερότητας όπως αυτή έχει εγγραφεί στη συνθήκη, αλλά ε, με προσοχή καταγράφουμε τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών όταν έχουν ανταγωνιστική δράση στην αγορά και δει σχέση με δυτικέ επιχειρήσεις πάλι με βάση τους κανόνες για τον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βιετναμέζοι φίλοι έχουν δεχθεί τη φιλοσοφία αυτή. Οι διαπραγματεύσεις όπως ήταν αναμενόμενο αποδεικνύονται περιπλοκές λόγω και της μεγάλης διάχυσης αυτών των ε, κρατικών επιχειρήσεων στο κρατικό σύστημα του Βιετνάμ. Από την άλλη είμαι ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλά αποτελέσματα και στο με αυτό. Εν γέννη έχουμε ολοκληρώσει 7 από τα 15 κεφάλαια για το εμπόριο και τη ε, τους δασμούς του εμπόριου, του εμπορίου, δασμούς, ε, συνεργασία γενική, ε, ανταγωνισμός, αντιμετώπιση των ε, trust, διαφάνεια και διαφθορά, σε σχέση με τις θεσμολογικές προτιμήσεις. Και εν τέλει, Πρόεδρε, όπως ξέρετε, ολοκληρώσαμε πρόσφατα μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συναλλαγών με το Βιετνάμ, που μεταξύ άλλων προβλέπει ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικές με τα όπλα μαζικής καταστροφής. Με βάση την κοινή προσέγγιση που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, σκοπεύουμε στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών να προβλέψουμε μια ρήτρα γέφυρα που θα συνδυάζει τις ρήτρες αυτές που έχουμε ενσωματώσει πριν από και το και το καιρό στα, κείμενά μας με το Βιετνάμ. Έχουν ξεκινήσει κάποιες συνομιλίες χωρίς να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Άρα δεν είναι ακόμη κομμάτι της συμφωνίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι της διαπραγμάτευσης με το Βιετνάμ και περιμένουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Όπω είπα, πολύ ευχαριστώ αν οι ε, κύριοι Βουλευτέ έχουν κάτι ακόμη να ρωτήσουν, να απαντήσω. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Πατρετσιόνε. Λάβαμε από την πρεσβεία του Βιετνάμ και ένα ενημερωτικό έγγραφο που τώρα μοιράζεται. Θα ακούσουμε τώρα τον πρέσβη. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη ε, της Επιτροπής. Ευχαριστώ τον ε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ε, για την εξαιρετική του παρουσίαση. Εγώ θα, θέλω να πω τα θα ήθελα να πω τα εξή. Οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία Βιετνάμ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν το 2012, τον Ιούνιο, ο στόχος μας είναι να είναι υψηλή ποιότητα και ολοκληρωμένη η διμερή συμφωνία για να τονώσει τις εμπορικές και γενικότερα οικονομικές σχέσεις των συμβαλωμένων μερών. Ε, φυσικά θα τηρηθούν οι κανόνες του ΠΟΕ και το εμπόριο στα αγαθά υπηρεσίες, οι επενδύσεις και άλλοι τομείς όπως τα, η προστασία των δικαιωμάτων διενετικής διατησίας, οι δημόσιες προμήθειες, η πολιτική ανταγωνισμού, ο βιωσιμός ανταγωνισμός και το εμπόριο θα ε, υπακούν στους αυτούς τους κανόνες. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ε, ε, που οφείλονται στα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και εκεί δημιουργούνται προβλήματα για την σταδιακή κατάργηση των δασμών ε, σε μια μεταβατική επταετή περίοδο από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να δοθεί κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά και ε, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τις επενδύσεις υπέρ, ε, πέρα από τις ε, δεσμεύσεις των συμβαλωμένων μερών στα πλαίσια του ΠΟΕ. Για δημόσιες προμήθειες διαπραγματευόμαστε για να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να δημιουργήσουμε νέες εμπορικές ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τους στόχους της δημόσιας πολιτικής αμφωτέρω των πλευρών η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ε, ε, διαφύλαξης προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η αμοιβαία αναγνώρισης και προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων ε, θα είναι γνώμονας και για τις δύο πλευρές στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, ήδη 11 γύροι έχουν γίνει και διάφορες ενδιάμεσες συσκέψεις. Έχουμε καταλήξει διάφορα επίπεδα συμφωνία για τους επιμέρους τομείς και έχουμε κλείσει κάποια από τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Στην τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού Βίντον Ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2014 ε, τονίστηκε και πάλι και από τις δύο πλευρές η σημασία της ε, ταχείας ε, σύναψης της συμφωνίας. Ε, ο κύριος Μπαρόσο, ο Πρωθυπουργός Γουίντεν Σούν και η Πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο να ολοκληρωθούν σε επόμενους μήνες οι διαπραγματεύσεις μετά τις οδηγίες που λάβαμε. Το Βιετνάμ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαπραγματεύσεων ω προ τα εκρεμή ζητήματα. Ένα εντατικό πρόγραμμα εργασία συμφωνήθηκε και ακολουθείται πλέον με απότερο στόχο να είναι φιλόδοξια η και ισόρροπη έκβαση των διαπραγματεύσεων όπως επιθυμούν και τα δύο μέρη. Μεταξύ άλλων ο στόχος είναι να αυξηθούν οι εμπειρικές συναλλαγές και ο ρόλος των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη να επικρατήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, να τεθούν σε ισχύ διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες. Είναι επίσης σημαντικό ε, να ισχύσει, ισχύσει η εγχώρη νομοθεσία για τα, την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων. Ε, για τα ε, δικαιώματα αυτά το Βιετνάμ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουμε βάσει της ισχύουσα συμφωνίας ώστε με αποτελεσματικότητα να εφαρμοστούν οι αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα βάσει των υποχρεώσεων μας που προκύπτουν από την δήλωση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την προστασία των ε, βασικών δικαιωμάτων. Έχουμε κυρώσει τις βασικές συμβάσεις του ILO και του ΔΟΕ και Ε, συνεχίζει τη διαδικασία για την ε, κύρωση ε, των υπολείπων. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε την συνεργασία με την Κίνα για αυτό το ζήτημα, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι άλλος ένας τομέας όπου επιθυμούμε και τα δύο μέρη να σημειωθεί η πρόοδος Ε, υπάρχει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, ε, εκπαιδευτικές ε, δραστηριότητες, δραστηριότητες κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αγνωσμένα εργαλεία όπως τις κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ για τις πολυεθνικές, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, η τριμερής δήλωση του ΔΟΕ για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική τους πολιτική. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί λοιπόν, αλλά υπολείπεται έργο το ώστε να μπορέσει να συναθεί η συμφωνία κατοχυρώνοντας τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα που θα είναι υποφελή και για τους, ε, τα άτομα και για τις επιχειρήσεις. Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει ε, βεβαίω ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Βιετνάμ και να επισύρει μια θετική πρόοδο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του Βιετνάμ. Επίσης θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη σημερινή ευκαιρία για να σας ζητήσω να στηρίξετε ε, την αναπτυσσόμενη χώρα που είναι το Βιετνάμ στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτή η συμφωνία έχει ιδιαίτερο βάρος για μας. Σας ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στα μέλη, και κυρίως τον συγητή μας εκ μέρους Επιτροπής να σας πω ότι προετοιμάζεται μια αντιπροσωπεία από την Διεθνή Επιτροπή Εμπορίου αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στη δεύτερη εβδομάδα του Απρίλη. Να ζητήσω τον κύριο Πετριτσόνε να ζητήσει από την Επιτροπή να ενημερωθεί για αυτό που είπαμε σήμερα. όπου ακούσαμε πολύ σημαντικές ε, πληροφορίες ενώ της επισκεψή μας στο Βιετνάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σαουρντήλ, ε, ο πρόεδρος μας. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε κύριε Πεσβευτά. Καλώς ορίζω και τον ε, επικεφαλή διαπραγματευτή μας. Θα είμαι σύντομος επειδή δεν έχουμε χρόνο και θα θέλω να αφήσω στους άλλους χρόνο για ρωταπαντήσεις. Αυτή η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο αν διεξαχθεί επιτυχώς για άλλες χώρες της Ασίας. Επίσης, από οικονομική σκοπιά, να σας υπενθυμίσω ότι τουλάχιστον δύο τρίτα του συνόλου των εξαγωγών του Βιετνάμ προέρχονται από τέσσερι μεταπητικέ βιομηχανίε. Εξάλλου, η ΕΕ παραμένει ο δεύτερο, μεγαλύτερο οικονομικό εταίρο για το Βιετνάμ, οπότε υπάρχει αμοιβαίο όφελο για τη συμφωνία αυτή που παρακολουθούμε προσεκτικά από την ομάδα παρακολούθησης. Θα συνεχίσουμε να το πράγμα αυτό όπως μας ενημέρωσε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων είχαμε σημαντικές επιτυχίες σε πολλά ζητήματα ιδιαίτερα όσον αφορά τους δασμούς, υπηρεσίες ε, συναλλαγών και άλλα Βεβαίω προς το τέλος των διαπραγματεύσεων παραμένουν τα πιο ακαθόδη αλλά έτσι γίνεται συνήθως να κάνουμε. Τα δύσκολα μένουν για το τέλος. Εγώ πάντως αισιοδοξώ και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων για το πρώτο δηλαδή του τρεχόντος έτους και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επικύρωσης στη συνέχεια. Έχουμε πολλές σημαντικές ημερομηνίες φέτος που σηματοδοτούν αυτή τη διαδρομή αυτών των επιτυχών διαπραγματεύσεων. Έχουμε και την ε, επέτειο επανένωσης του Βιετνάμ που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία. Το Βιετνάμ βεβαίως είναι έτσι φιλόδοξο επειδή διεξάγει διαπραγματεύσεις εμπορικές και με άλλους άλλους χώρες του ειρηνικού και προετοιμάζεται να προσυπογράψει μια συμφωνία εμπορική με τη Ρωσία. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε γρήγορα και με επιτυχία. Εδώ θα σταματήσω πάντως. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας από την ομάδα παρακολούθησης. Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά αυτές τις τελευταίες φάσεις της διαπραγμάτευσης και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευτεί επιτυχώς παρά τα λίγα τελευταία ακαθόδη ζητήματα. Νομίζω θα επιτευχθεί επιτυχία. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρέφομαι προς τους Σκιώδης. Φρανκ Α, από το ΕΛΚ. Έχεις το λόγο Φρανκ. Ναι, Πρόεδρε. Χαιρετώ τον πρέσβη και το εκφράζω την χαρά μας που τον υποδεχόμαστε εδώ και του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του διαπιστώνουμε όλοι τη δουλειά που έχει γίνει σωστά από τον διαπραγματευτή μας που χαιρετίζω επίσης. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία με λίγα τελευταία ζητήματα προς επίλυση, όπως είπε και ο προλογής σας, τα πιο καθόδη. Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα για το δεύτερο ήμιση του 2015. Εμείς το επιθυμούμε αυτό, γιατί μας φαίνεται σημαντική η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Δύο ζητήματα πάντως να αναφέρω για τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή. Καταρχάς, οι άδειε για τα εινοπνευματόδη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς στο Βιετνάμ από το 2013 που έχει κινδύνους για την διανομή και την πώληση υνοπνευματοδών ποτών. Οπότε τι γίνεται εκεί, ποια είναι τα αποτελέσματα και θα ήθελα να μάθω επίσης αν η βιετναμική κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεύτερο ζήτημα, φυτογενομικός έλεγχος υπάρχουν επαρκείς εγγυήσει για τον υγειονομικό και φυτο-υγειονομικό έλεγχο σχετικά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πολλοί κλάδες της οικονομίας της δικής μας ε, έχουν έρθει μαζί μας για αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα από τις ιδιοκαλλιεργίες και άλλους τομείς. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν κάτι γι' αυτό. θα πάω και εγώ με την Ίντα 6 με 10 Απρίλη στο Βιετνάμ και θα ήταν βεβαίω να δούμε τα συμπεράσματα αυτή εδώ τη συνεδρίαση και του μελλοντικού γύρου στο Βιετνάμ. Πάντω με χαρά θα ταξιδέψουμε για να σα ακούσουμε και θα θέλαμε βεβαίω να ολοκληρωθεί σύντομα η συμφωνία αυτή που ξαναλέω είναι πολύ σημαντική στα πλαίσια των εμπορικών μα συναλλαγών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ναι, ευχαριστώ και εγώ τον, τον πρεσβευτή και τον διαπραγματευτή για την παρουσίαση που κατέδειξε την σημασία της συμφωνίας αυτής καθεαυτής ως πιθανό μοντέλο και για άλλες χώρες. Έχω δύο γρήγορα ζητηματάκια. Δεν έχουμε χρόνο να τα πω γρήγορα. Πρώτον, ο συσχετισμός της διαπραγμάτευσης αυτής με την άλλη διαπραγμάτευση στην οποία συμμετέχει αυτή τη στιγμή το Βιετνάμ. Στα πλαίσια του TTIP. Και για τα χρονοδιαγράμματα της διαπραγμάτευσης επειδή ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται πολύ οι Αμερικανοί για αυτές τις διαπραγματεύσεις Οπότε διαρωτούμαστε κατά πόσο αυτό επηρεάζει την επιβράδυση των πραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενό και αφετέρου για το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε. Γιατί ξέρουμε ότι και πάλι εδώ υπάρχει πίεση από τη ΣΥΠΑ, ώστε κάποια κεφάλαια να μοιάζουν περισσότερο με αυτό που αρέσει στους Αμερικανούς και για τα οποία εμείς έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία IPR και γεωγραφικές ενδείξεις. Δεύτερη ερώτηση ευαίσθητα προϊόντα που αναφέρθηκαν. Για την Ευρώπη νομίζω είναι βεβαίως κρίσιμη σημασία η πλήρης, ε, το, πλήρη, το πλήρες άνοιγμα αγοράς κάποιων προϊόντων όπως το ρύζι για τα, για τα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Οπότε ρωτάω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζεται ώστε να καταστήσετε έτσι βαθμιαία αυτό το πλήρες άνοιγμα της αγοράς, ιδιαίτερα σε τόσο κρίσιμα προϊόντα όπως το ρύζι. Τελευταία ερώτηση, δημόσιοι διαγωνισμοί. Από τις συζητήσεις και τα κείμενα που είδαμε, γνωρίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε κυρίως με ένα άνοιγμα των διαγωνισμών για τις δύο αστικές περιοχές Ανόη και Χότσιμίν, οπότε Ισχύει αυτό ακόμα, ρωτάω. Ή μήπω έχετε προβλέψει μια βαθμιά έτσι, επέκταση και στην υπόλοιπη χώρα. Αυτά από μένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάκη. Άλτε. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ. Θέλω να ορίσω τον Πρεσβευτή και του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μαρία Ντεσόρνη είναι η ε, πρόσωπο τη ομάδα. Οι διαπραγματεύσει με το Βιετνάμ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο τέλο του έτου, όπω ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε να καταλήξουν σε μια συμφωνία καλή για όλου. σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Θέλουμε μη ιδεότητα σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά του Βιετνάμ, καλύτερη αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων προέλευσεως, ιδιαίτερα για τα προϊόντα κρασιού και αλκοόλου και κανόνες προελεύσεως επίσης. Για την επικύρωση της ε, εμπορικής συμφωνίας θέλουμε μια φιλόδοξη και καλή συμφωνία. Προς και των δύο λαών. Το Βιετνάμ αναπτύσσει την οικονομία του με ρυθμούς ανάπτυξη 5% όπως μας λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι όμως ακόμα αναπτυσσόμενη χώρα και κάθε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο το εμπόριο και το λόγο. Δεν πρέπει βέβαια αυτά να γίνουν εις βάρος της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Είναι αυτά θέματα τα οποία πρέπει να μπουν στο κεφάλαιο της βιώσιμης αλλά τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την εφαρμογή τους. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή της συμφωνίας και τα θέματα των συμφωνών δικαιωμάτων τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ιδέα θα ήταν να αποσταλούν για το διάλογο για τα θέματα δικαιώματα παρατηρητέ από πλευρά μα. Επίση θέλουμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή πώ σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των δικαιωμάτων και να προστατεύσει τα θέματα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Έχουμε δε ένα θέμα που αφορά προσφυγή οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με κυβερνητικών οργανώσεων, δύο τον αριθμό των τον Ombudsman, εις βάρος της Επιτροπής για την τρόπο που θα χειριστεί σχετικά θέματα. Και πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Να ευχαριστώ. Γκουα, δεν έχετε παρατηρήσεις. Πράσινη. Ροντρίγκες. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πρεσβευτή και τον διαπραγματευτή για την παρουσία τους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Να επιθυμίσω ότι οι σχέσεις της Ένωσης με το Βιετνάμ ενισχύθηκαν από το 1995 όταν υπό Ισπανική Προεδρία υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία συνεργασία μεταξύ ΕΕ Βιετνάμ. Και ιδιαίτερα το Βιετνάμ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα εθνικά ή και περιφερειακά προϊόντα από τη δικιά μου χώρα. Κλώς το υφαντουργικά, υποδήματα, ρύζι και κεραμική να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η κυρία Μόσκα στις ερωτήσεις της προς την Κομισιόν. Τι μέτρα θεωθετήσετε για τα ιδιαίτερα βάλωτα προϊόντα τα οποία θα εκτεθούν στο πλήρες άνοιγμα των αγορών. Τι γίνεται λοιπόν με την εξισορρόπηση, τη σωστή εξισορρόπηση των επιπτώσεων της συμφωνίας για αυτά τα προϊόντα. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μας πει αν θα μπορούσε στην ιστοσελίδα της να αναφέρει περισσότερα για τα αποτελέσματα του κάθε γύρου διαπραγματεύσεων. Πρέπει να έχουμε όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται για αυτό το θέμα και να πω προς τον κύριο Πρεσβευτή το εξής. Δύο ερωτήσεις τι φιλοδοξία έχει η κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα του Βιετνάμ σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, με την Ένωση. Δεύτερον, από την εμπειρία που έχουμε στις εμπορικές συμφωνίες και για το πώς εφαρμόζονται κάποιες στην πράξη, νομίζω ότι μια στρατηγική ανακοίνωσης που δεν διέρχεται μόνο από τη διάθεση των πληροφοριών αλλά από την κατάδειξη των πλεονεκτημάτων για όλα τα μέρη της συμφωνίας μικρομεσαίους του Βιετνάμ τους ομολογούς τους της Ένωσης και τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η νέα συμφωνία νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλέξουμε βέβαια σε μια συμφωνία σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονδιάγραμμα είναι σημαντικό να έχουμε καλή συμφωνία αλλά θα πρέπει όσο μπορούμε η συμφωνία αυτή να φτάνει και να εποφελεί όσο γίνεται περισσότερους. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και στο Βιετνάμ αλλά και στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μας υπενθυμίσατε σε όλους και στους συναδέλφους ότι τελειώνει ο χρόνος. Ερωτώ τους βουλευτές αν θέλουν άλλοι να λάβουν το λόγο. Ιδάλλως διατυπώθηκαν ερωτήσεις. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να πει η Επιτροπή και ο προσβευτής μετά. Κύριε Πετριτσόνα, εσείς πρώτα. Thank you very much, Chairman. I shall try and be brief and... Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Αν τυχόν ε, ξεχάσω κάτι, παραλείψω κάτι ή δεν σας δώσω αρκετές λεπτομέρειες, Ευχαριστώ ε, διμερώς ε, να συνεχίσουμε και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Για το μοντέλο των διαπραγματεύσεων, όπως είπε ο κ. Ζαραντήλ και άλλοι, λοιπόν θα απαντήσω αποφατικά Απολύτως ισχύει αυτό, δηλαδή το μοντέλο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς και για άλλες ε, συμφωνίες με άλλες χώρες. Με τη Σιγκαπούρη παραδείγματος χάρη που είναι η πλέον ε, αναπτυγμένη χώρα από τις μεγάλες χώρες του ΑΣΕΑΝ με το Βιετνάμ που είναι στην αντίθετη άκρη ως προς την ανάπτυξη. Είναι εντυπωσιακός αναπτυξιακός ρυθμός παρόλα αυτά το Βιετνάμ. Ε, νομίζω ότι έτσι θα ορίσουμε το πλαίσιο για την περιοχή Ασιαν. Περισσότερες διαπραγματεύσεις, ώστε ε, ε, ο απότερος στόχος να υλοποιηθεί, δηλαδή να συνάψουμε μια συμφωνία περιοχή προς περιοχή, region to region, σε, κατά τη διαστολή με μονομένες συμφωνίες. Θα δούμε τι είναι επωφελέστερο. Θα χρειαστεί χρόνο βεβαίω, αλλά θα συνεχίσει η διαδικασία. Η σχέση με το TBT είναι πολύ άπληστοι οι Βιετναμέζοι φίλοι μας. Θέλουν το ταχύτερο δυνατόν να συνάψουν τις δύο συμφωνίες και να αποκομίσουν το ωφέλη και από τις δύο. Ξέρω ότι έχουν ένα πρόβλημα ικανοτήτων. Νομίζω ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Βιετνάμ αποτελεί που ιδιαίτερη πίεση, αλλά το σταμάζουμε. Συνεχίζουν ε, με αμύωτο ρυθμό και τις δύο διαπραγματεύσεις. Ε, σε καμία περίπτωση δεν έχουν ε, αργότερο ρυθμό λόγω των διαπραγματεύσεων TPP και παρότι το περιμέναμε αυτό, γιατί το έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες περιπτώσεις όπου το δυναμικό είναι και μεγαλύτερο σε σχέση με το Βιετνάμ, εντυπωσιακό. Νομίζω ότι το Βιετνάμ έχει ε, μια ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το ρόλο που θα έχουν οι συμφωνίες για την αναπτυξιακή τη πολιτική και πορεία. Και στην προχωρά πολύ ε, στοχευμένα. Αναφερθήκαμε σε σημείο όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις. Νομίζω ότι στην συμφωνία με τον Καναδά αποδείξαμε πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να επιτύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας για γεωγραφικές ενδείξεις για τα προϊόντα μας, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε και περιφέρω ελιγμών στους εταίρους μας για να προστατεύσουν και εκείνοι τα εμπορικά τους συμφέροντα, τις εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες να μετάσχουν ε, σε διαπραγματεύσεις τύπου TPP όπου συμμετέχει και ο Καναδάς. Η Χιλή επίσης ε, συμμετέχει και ε, αυτές οι χώρες έχουν συστήματα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που είναι παρεμφερή με τα δικά μας δεν αμφιβάλλω ε, ότι μπορεί να επιτύχει ε, το, την ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα και το Βιετνάμ. Ευαίσθητα προϊόντα. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα για το πώς χειριζόμαστε τα ευαίσθητα ζητήματα. Ρύζι είναι καταφανώς ένα ευαίσθητο προϊόν. Δεν ε, φαίνεται πιθανία η απελευθέρωση του εμπορίου όμως, σε αυτόν τον τομέα, όμως μπορούμε να έχουμε δασμολογικές ποσοστώσεις, τέτοιου τύπου εμπορικά εργαλεία ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε κάποια όρια, ανώτατα όρια για να ελέγχουμε την, ε, ε, τον αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά. Το Βιετνάμ είναι πολύ σημαντικό στους εξαγωγές ρυζιού και θα πρέπει να, βρούμε, να βρεθεί μια ε, συμβαστική λύση διότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι ευαίσθητο το προϊόν για το Βιετνάμ και πρέπει ε, κάποιος ε, να αναρωτηθεί ότι αν δεν γίνει σεβαστό αυτό ποιο είναι και το όφελος για το Βιετνάμ να συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Τώρα βοηδή, και, ε, βοηδές και χείριο κρέας με τον Καναδά, στη συμφωνία με τον Καναδά και εκεί πάλι καταλήξαμε σε μια ισορροπία που μπορεί να μην ήταν τέλεια αλλά έγινε αποδεκτή από, το, από όλους Για τα κλωστοϊφαντοργικά διαφέρει η κατάσταση. Ε, είναι διατεθειμένοι να δεχθούν την άνευ πρόσβαση στην αγορά και μπορώ να σας πω επίσημα ότι το Βιετνάμ δεν πρόκειται να προβάλλει αντιρρήσεις ε, για την εισαγωγή βιετναμέζικων προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το καθώς προέλευσης θα είναι ε, καταλητική σημασία της διαπραγματεύσεις. Λύση δεν έχουμε βρει ακόμη. Το Βιετνάμ νομίζω έχει κάνει ε, πολλά βήματα τη διπλή ε, μεταποίηση για τον ε, καθεστώς προέλευσης το έχει δεχτεί ήδη το Βιετνάμ και έτσι η κλωστοφοντολογική βιομηχανία του Βιετνάμ μπορεί να αυτομεταρρυθμιστεί και να απομακρυνθεί από την υπερβολική εξάρτηση από τις εισαγωγές από την Κίνα. Δεν είναι απλή η διαπραγμάτευση. Θα είναι ένα από τα τελευταία ζητήματα που θα ρυθμίσουμε Υπάρχει όμως μεγάλη αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές για να εξευρεθεί λύση. Για τις οικοάδειες αυτό χρονολογείται από την προσχώρηση του Βιετνάμ στον ΠΟΕ. Δεν προτιθέμεθα να επαναδιαπραγματευτούμε ε, δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί ήδη από το Βιετνάμ στα πλαίσια του ΠΟΕ Ζητούμε από το Βιετνάμ να τροποποιήσουν το καθεστώς ώστε να τηρήσουν, εκπληρώσουν ε, τις δεσμεύσεις τους και να μην παρεμποδίσουν την πρόσβασή μας για αυτό το προϊόν. Φυσικά νομοποιούνται και ανησυχίες που έχει το Βιετνάμ για, για το, τα θέματα απάτης, ε, τα φορολογικά ζητήματα, για όλα αυτά τα προϊόντα όμως. Ξεκολουθούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να παρεμποδιστεί το εμπόριο. Ε, είναι ένα θέμα που φροντίζουμε να εξετάζουμε ε, συστηματικά. Για τα φυτογενομικά ε, πρότυπα η πολιτική μας είναι ότι δεν ε, διαπραγματευόμαστε φυτογενομικά μέτρα στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Αυτό που διαπραγματευόμαστε είναι όρους, εφαρμοστικούς όρους για τα φυτογενομικά μέτρα σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΠΟΕ. Τώρα, ε, η οικονομική κατάσταση της χώρας, η νομοτεχνική ικανότητα του Βιετνάμ για τη διαχείριση αυτών των διατάξεων είναι θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, έχουμε εξετάσει το θέμα της τεχνικής αρρωγής προς το Βιετνάμ σε αυτό το τομέα και θα συνεχίσουμε τα βήματα που έχουμε κάνει αναφυσβήτητα. Δεν πρόκειται να τροποποιηθούν τα φυτογενομικά μέτρα μας. Για τις δημόσιες ε, συμβάσεις, τις δημόσιες προμήθειες, διαπραγματευόμαστε τις δύο δεσμεύσεις σε εθνικό επίπεδο, ε, στην περίπτωση του Καναδά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καλά βαίνουν οι διαπραγματεύσει, δεν είμαστε 100% ικανοποιημένοι, όμω θα εφαρμοστούν σε όλο το Βιετνάμ ε, τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα σε υποεθνικό επίπεδο προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε διότι ανατίθεται δημόσια προμήθειες σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο και το Βιετνάμ για το Χανόι και το Μίνθα δείχνει ευελιξία. Ε, και επιθυμούμε να διευρυνθεί η κάλυψη και σε άλλες περιοχές αλλά ε, συνεχίζονται ακόμη οι διαπραγματεύσεις, δεν έχουμε καταλήξει τέλος. Ανθρώπινα δικαιώματα και αποτίμηση, αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση της πολιτικής και των διαφόρων πτυχών των σχέσεων μας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το μέρος όπου έχει σημειωθεί ε, σταδιακά πρόοδος. Στη διαπραγματευτική μας εντολή την αρχική για το Βιετνάμ δεν προβλεπόταν να κάνουμε εξποστα αξιολόγηση αντικτύπου. Ταυτόχρονα είναι πηγή σημαντικής ανησυχίας ε, στο Κοινοβούλιο, στην Κοινωνία των Πολιτών, στα κράτη-μέλη τέτοια ζητήματα και τώρα με την Επιτρόπο ε, Μάλμστρομ συζητούμε για να βρούμε τρόπους να εστιάσουμε την προσοχή μας στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Βιετνάμ. Έχουμε ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία. Θα έχουμε και μια ρήτρα σύνδεση με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Έχουμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα δούμε ποια άλλα εργαλεία μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να συνεχίσουμε να συνδράμουμε το Βιετνάμ ως προς την μεταξέλιξη κατάσταση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, ε, δημόσια πληροφόρηση, ε, πρόσβαση στα έγγραφα. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει τις τακτικές εκθέσεις που υποβάλλουμε μετά τους γύρους των διαπραγματεύσεων. Την ίδια έκθεση στέλνουμε και στα κράτη-μέλη. είναι μια επίκαιρη και ακριβής έκθεση κατά τη δική μας αντίληψη ε, μετά την ολοκλήρωση κάθε διαπραγματευτικού γύρου με χαρά να ε, προσκομίσουμε στοιχεία ε, στο Κοινοβούλιο μετά το, την αποστολή μας τον Απρίλιο στο το Βιετνάμ και μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία μας για να εξυπηρετηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Σας ευχαριστούμε. Στρέφομαι και πάλι σε εσά, πρέσβη. Ε, ίσως μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις σε σχέση με τις ερωτήσεις που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ορισμένες είναι πολύ καλές και ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει απαντήσει περισσότερες από τις ερωτήσεις ε, Ωστόσο, θα ήθελα σε ορισμένα σημεία να δώσω ιδιαίτερη έμφαση. Καταρχά, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σα πω ότι το Βιετνάμ πραγματεύεται συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών μια σειρά από εταίρου, όπω σημείωσε και ο κύριο Σαχάντιλ. Θα ήθελα ιδιαίτερα να πω ότι στι ε, συμφωνίε που έχουμε αντίστοιχα με τι ΗΠΑ και άλλου εταίρου είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή, στην ολοκλήρωση των δεδομάτων και την υπογραφή και αντίστοιχα προχωρούμε σε ολοκλήρωση συναλλαγών με πολύ μεγάλους εταίρους όπως είναι η Κορέα, πολύ μεγάλος εμπορικό εταίρος για το Βιετνάμ τις σχετικέ διαπραγματεύσεις ολοκληρώσαμε στις τέλος του 2014 με τη Ρωσία, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία επίσης έχουμε προχωρήσει σε άρσεις των τελωνιακών, των δεσμολογικών ε, επιβαρύνσεων με την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία και με άλλους εταίρους επίσης. Και έτσι τώρα ιδιαίτερα προχωρούμε στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν εμπειρία από διαπραγματεύσει με σημαντικού εταίρου εκ μέρου του Βιετνάμ. Παράλληλα, συνεχίζουμε διαπραγματεύσει με μια σειρά από χώρε. Και πιστεύουμε ότι μπορεί ένα εταίρο να μα βοηθήσει στη διαπραγματεύσει με άλλου εταίρου. Στι χώρε ΕΑΝ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ολοκληρωμένε ε, συμφωνίε μόνο με τη Σιγκαπούρη από τι χώρε ΑΣΕΑΝ. Είναι, είναι πιο ανεπτυγμένη από τι χώρε ΑΣΕΑΝ η Σιγκαπούρη. Όμω η δεύτερη σε ανάπτυξη είναι το Βιετνάμ. Γι' αυτό και υπογραμμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο το Βιετνάμ για πολλέ χώρε του κόσμου. Και ιδιαίτερα προωθεί τις απρόσκοπτες συναλλαγέ στην παγκόσμια οικονομία. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση την θεωρούμε πάντα ως έναν από του πιο σημαντικού εμπορικού εταίρους του Βιετνάμ. Ο εμπορικός όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών πέρυσι ήταν 35 με 36 δισεκατομμύρια. Και δεν θεωρούμε, εάν τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία, να αυξηθεί κατέτος κατά, τα, κατά ένα ποσοστό 15 με 20% ο όγκος αυτός. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμεί να δει ο λαός, οι επιχειρήσεις το κράτος του Βιετνάμ. Θέλουμε να το δούμε και γι' αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε και την και θέλουμε να διατηρήσουμε ταυτόχρονα και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη του Βιετνάμ με στόχο 6% ανάπτυξη το χρόνο. Το 2014 είχαμε ε, ανάπτυξη 6% στην οικονομία του Βιετνάμ παρά τις δυσκολίες που οδήγησαν σε μια επιβράδυνση στην οικονομία και δυσκολίες εσωτερικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εταίρος για τις εξαγωγές του Βιετνάμ. Όμως ε, πέρσι ήδη υπερκαλύφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα τώρα για, την αγορά του Βιετνάμ, την εξαγωγική αγορά του Βιετνάμ, είναι πλέον δεύτερη σε σειρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είναι καλή ε, και σκόπιμη μια Συμφωνία των Συναλλαγών, Όπω και να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του κύριου εταίρου του Βιετνάμ. Για κάποια ιδιαίτερα ζητήματα που ζήτησαν περισσότερε πληροφορίε οι βουλευτέ κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση, Θα ήθελα να αναφερθώ στις αποφάσεις που έχουν συζητηθεί ευρέως μεταξύ των πολιτών, γιατί ξέρετε εμείς στο Βιετνάμ για τα θέματα της κατανάλωσης του αλκοολούχων προϊόντων. Ξέρετε, εμείς έχουμε μεγάλη παράδοση. Είμαστε η τέταρτη μεταξύ των χωρών του ΑΣΕΑΝ στην κατανάλωση αλκοόλ. Τρία δις ευρώ το χρόνο πηγαίνουν μόνο στην κατανάλωση της μπύρας. Αν επισκεφθεί κανείς το Βιετνάμ θα διαπιστώσει ότι υπάρχει κάθε τύπου και μάρκα μάρκας μπύρα. Βελγική θέλετε, γερμανική θέλετε, από οπουδήποτε στον κόσμο θα βρείτε μπύρες. Το αλκοόλ λοιπόν είναι και ένας από τους κύριους λόγους τροχαίων ατυχημάτων. Μόλις τώρα εορτάσαμε τον, ε, το νέο έτος, το συλληνιακό νέο έτος και ο αριθμός των τροχαίων που οφείλονται σε ένα βαθμό στην κατανάλωση του αλκοόλ έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. Στις εννέα ημέρες που κρατάνε που κρατάει η αργία για το νέο έτος, είχαμε πάνω από 300 νεκρούς σε τροχέα, τα οποία σε ένα βαθμό οφείλονται, σε ένα βαθμό υπογραμμίζω, στην κατανάλωση του αλκοόλ. Άρα το θέμα των αλκοολούχων ποτών και η σχετική επαφή έχει στηθεί πολύ και στην κοινή γνώμη και στην κυβέρνηση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπε και ο κύριος ότι υπάρχει αιτητική συνομιλία για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε και με πολλές άλλες χώρες, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλες χώρες. Η κατάσταση σχετική με τα δικαιώματα στη χώρα μας έχει βελτιωθεί καθέτος, όπως αναγνωρίζουν και οι διεθνείς οργανώσεις. Πρόσφατα δε, στα τέλη του Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε μάλλον ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επί τη ευκαιρία δε ταξιδιού μια αποστολή μα στι Βρυξέλλε, πέρασαν και από το Βερολίνο για να επισκεφθούν μια φυλακή στο Βερολίνο, ώστε να σωματωθεί και αυτή η εμπειρία στι συνομιλίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και αυτό τον διάλογο. Βεβαίω και πρέπει να ενισχυθεί, όπω είπατε και εσεί, η ευαισθητοποίηση των ε, ε, πολιτών σε σχέση με, τις ε, με τα δυνάμει ωφέλη μιας της συμφωνίας για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες εκατέρωθαν, αλλά πάνω απ' όλα στο Βιετνάμ. Έχουμε πλήρη συνέντευξη της σημασίας και ιδιαίτερα καταβάλουμε προσπάθειες για να καθιστούμε δημόσια και να διαφημίσουμε όπως είναι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε πολίτες αλλά πάνω από όλα να ενημερώνονται και να προετοιμάζονται για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι τελευταίες δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι δεν είναι ενήμεροι οι επιχειρηματίες για τις διαπραγματεύσεις ή για την πρόοδο αυτών και τις συνέπειές τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας ε, απασχολήσει ιδιαίτερα η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση. Και πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να τις καλέσουμε να προετοιμαστούν όχι μόνο για τις μεγάλες ευκαιρίες αλλά και για τις προκλήσεις που θα φέρει η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών που διπραγματευόμαστε με άλλους εταίρους. Και θα ήθελα και εσάς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμφωνήσετε, να σας παρακαλέσω να συμφωνήσετε ώστε να εξασφαλιστεί υποστήριξη του Βιετνάμου τι όμενε χώρες γιατί όπως είπα έχει πολύ μεγάλη σημασία η εταιρική σχέση του Βιετνάμ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην δουλειά σας ολοκληρώνοντας ο συγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους Κιώδης για την δέσμευση και την συμμετοχή τους, την εργό. Ευχαριστώ και τους αδέλφους που πήραμε εδώ στη συζήτηση. Ευχαριστώ τον επικεφαλή των διαπραγματεύσεων και την ομάδα του για τη δουλειά που έκαναν και ευχαριστώ και την εξοχότητά του κύριο Πρεσβευτή γιατί στην προηγούμενη του θητεία ήταν στη χώρα μου και έχουμε έτσι κοινέ αναμνήσεις από την παρουσία του στην Τσεχία. Αυτά από μένα και με χαρά θα συνεχίσω τη δουλειά μα στην ομάδα παρακολούθηση για τον μέλλον των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανακοίνωση μετά από αυτό το σημείο. Έχουμε ακόμα 40 λεπτά και δύο σημεία στην ημερήσια. Αν θεωρείτε ότι μπορούμε να τελειώσουμε το τελευταίο σημείο 40 λεπτά, εντάξει, αλλιώ το αναβάλουμε. 17 στην ημερησία. Εξωτερικές επιπτώσεις του εμπορίου σε χώρες εκτός ΕΕ. Πρώτη αλλαγή απόψεων έχουμε τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, τον εισηγητή του κ. Ζαχάντιλ. Από ό,τι καταλαβαίνω αποβλέπει στο να διαφωτίσει τις σχέσεις μας τις εταιρικές με ιδιώτες σε τρίτες χώρες. Θα δίνω το λόγο στην εισηγητή παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Λαμβάνω σοβαρά αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε χρόνο, έχουμε δύο σημεία και μόνο 40 λεπτά. Θα είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται. Εδώ έχουμε ένα πρώτο έγγραφο εργασία που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία που ονομάζουμε Εξωτερικό Αντίκτυπο του, της πολιτικής εμπορίου Ε, στις πρωτοβουλίες των χώρες εκτός Ένωσης. Δηλαδή με άλλα λόγια προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες των προγραμμάτων ΣΔΙΤ και προσπαθούμε να εμπλέξουμε τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ένωση σε οικονομικέ δραστηριότητες εκτός αγορών Ένωσης. Χωρίζεται το έγγραφο σε έξι τμήματα. Έξι κύρια τμήματα. Που βεβαίω δεν χρειάζεται να καθορίσουμε αυτό το PPP γιατί όλοι γνωρίζουν τον ορισμό του θέματος αυτού Νομίζω ότι αποδεχόμαστε τη διαδικασία αυτή. Παρ' αυτά σε κάποιες αγορές αναπτυσσόμενες εκτός ένωσης είναι αρκετά χρήσιμο να υπάρχει συμμετοχή ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και να υπάρχει διείσδυση στην οικονομική δραστηριότητα αυτών των χωρών τώρα, όπως λέει σε μία παράγραφο στη δεύτερη συγκεκριμένα για την δημιουργία υποδομών ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών σε κοινοφιλείς επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές επιχειρήσεις κλπ. Να τονίσω ότι εστιάζομαι κυρίως στις αμπτυσσόμενες αγορές σε χώρες εκτός Ένωσης όπου το επίπεδο ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή η διαφορά και η έλλειψη δημοσίων υποδομών αυξάνεται. Μπορούμε να δούμε λοιπόν σε αυτές τις χώρες να υπάρχει έλλειψη βασικών υποδομών από όλες τις απόψεις και τα ΣΔΙΤ θα μπορούσαν βεβαίω να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την βελτίωση των υποδομών. Στο σημείο 3 έχουμε επίσης μια περιγραφή συγκεκριμένων χωρών που είναι ιδιαίτερα ενεργές στην πρόθεση αυτό το σχεδίο. Και γίνεται αναφορά σε οργανώσεις, σε συμφωνίες, συνθήκες και προγράμματα που προωθούν αυτή τη δικασία. Στο σημείο 4, τα κριτήρια και οι αρχές. Έχουμε μια προσπάθεια δηλαδή να χωρίσουμε αυτό το μας σε δύο κατηγορίες, έτσι, ευρείς κατηγορίες το θεσμικό ΣΔΙΤ, PPP, και το PPP που αφορά τις συμβάσεις, ανάλογα με το πώς συνάπτονται και πώς χρηματοδοτούνται. Έχουμε επίσης και πιο λεπτομερείς αναφορές για διάφορα είδη αυτών των σχέσεων, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν, όπως περιέγραψα. Θα βρείτε επίσης εδώ και μια δέσμη βασικών κανόνων, αρχών, που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν στα πλαίσια του PPP. Διαφάνεια, σχεδιασμός, value for money, σημαντική εμπλοκή των stakeholders και λογοδοσία. Επίσης, το πιο σημαντικό εδώ είναι το σημείο 5 στο αρχικό σχέδιο κειμένου και στο σημείο 6 επίσης όπου θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή για το πώς γίνεται η εφαρμογή των σχεδίων PPP εκτός Ένωσης και δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρέχουν νέες ευκαιρίες για τις νέες επιχειρήσεις ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες. Επίσης, θα δείτε και τις προκλήσεις εδώ να αναφέρονται από συγκεκριμένα, συγκεκριμένα σχέδια. Πάντως να υπογραμμίσω ότι δεν προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγές στην εσωτερική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα νομικά πλαίσια. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Απλά και μόνο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα πλαίσια για την καλύτερη προώθηση της λύσης PPP ή του σχεδίου των εγχειρημάτων PPP στις αγορές εκτός Ένωσης. Θα βρείτε εδώ μια περιγραφή αυτών των προκλήσεων στη συνέχεια του κειμένου πιο κάτω. Νομίζω αυτά από μένα. Θα είχα να σας πω. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση. Και θα μπορέσουμε ελπίζω να συσχετίσουμε το χείρημα αυτό με άλλε κοινωνικέ πολιτικέ, πολιτικέ που αφορούν την ανάπτυξη και τι δραστηριότητε ανάπτυξη τη ΕΕ σε τρίτε χώρε. Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτησή μα και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια αμοιβαία συμφωνία που θα μας βοηθήσει να συντάξουμε μια αποδεκτή και θετική έκθεση πρωτοβουλία στο τέλος. Αυτά που με ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συζητάμε εδώ πέρα τις εντοχές συμβάσεις ε, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών. Έχουμε τους stakeholders, έχουμε την κυρία Κένιχελ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την υπηρεσία της χρηματοδότησης των PPP. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχω φτιάξει μια παρουσίαση, θα σας τη στείλω με email για να την έχετε. Έχω κάνει κάποια αντίτυπα. Θα είμαι σύντομη πάντως και θα μιλήσω μόνο για κάποια βασικά σημεία που προετοίμασα. Η ΣΔΙΤ ε, είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το λένε και περισσότερο σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, διότι είναι, αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματικός μηχανισμός ε, για την παροχή βασικών υπηρεσιών στους υποδομές. Έχουν γίνει κάποιες εκτιμήσεις ε, ότι ε, η ανάγκη που δεν καλύπτεται για ε, τη χρηματοδότηση των υποδομών σε αναπτυσσόμενες χώρες ανέρχεται σε ένα τρεις το χρόνο. Είναι δυσθεώρητο το ποσό και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το χάσμα για να το καλύψουμε με εθνικούς προϋπολογισμούς εις ΣΔΙΤ Μπορεί να είναι ένας τρόπος ε, για να ενισχύσουμε τη νέα γενιά ε, υποδομών ε, που απαιτούνται πέρα από αυτά που μπορεί να χρηματοδοτήσει κάθε κράτος. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν πολλές χώρες αναπτύξει ε, της ΔΙΤ, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία είναι οι πρωταθλητές ε, στον τομέα των ΣΔΙΤ ε, ε, στην Κίνα και στη Βραζιλία και την Τουρκία πολλές εταιρείε φτιάχνουν, επιχειρούν σδίτες στην χώρια αγορά και οι σημαντικότεροι επενδυτές στην Αλοδαπή είναι και πάλι η Τουρκία αλλά και η Ισπανία και η Κίνα. Γιατί στρέφονται οι χώρες σε αυτό το εργαλείο. Ε, για να απελευθερέσουν ε, πόρους, κονδύλια, όπως έλεγα, για να επισπέσουν την ε, κατασκευή υποδομών. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε αυτό για την ίδρευση, υδροδότηση για την, τις οδικές υποδομές. Χρειάζεται υπερβολικά πολλής χρόνος για να χρηματοδοτηθεί αυτό με δημόσια κονδύλια και έτσι βρίσκουν promoters, ε, φορείς που αναλαμβάνουν ε, την, ε, τα, τα προγράμματα για τις υποδομές. Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το έγγραφο εργασίας σας που είναι παρεμπιπτόντως πολύ καλογραμμένο ε, και διαπίστωσα ότι δεν αναφέρεστε σε ορισμό. Εμείς στην ΕΤΕ θεωρούμε ότι ορίζεται η ΣΔΙΤΜΗ ως συμβατική σχέση ανάμεσα σε ένα δημόσιο και ιδιωτικό ε, φορέα ανάθεσης, ο οποίος θα παράσχει δημόσιες υπηρεσίες ε, σε ένα τομέα βασικών υποδομών και θα συμφωνήσει να έχει ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο αποτέλεσμα και γι' αυτό βάσει της απόδοσης θα αποζημιωθεί. Για να ξέρουμε ε, τι στείτε και τι χρειάζεται από πλευράς του κράτους, χρειάζεται διαγωνισμός, ανταγωνιστική διαδικασία, τους ώστε να ευρεθεί ο φορέας που με το χαμηλότερο δυνατό κόστος θα ε, έχει τις καλότερες παροχές. Επίσης χρειάζεται μια αρχικά υψηλή επένδυση, μην το ξεχνάμε, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό προκαταβολικά, να αναλάβει προκαταβολικά μεγάλο μέρος του κινδύνου προτού αποζημιωθεί από το δημόσιο τομέα. Αυτά προβλέπονται στη συμβατική σχέση ανάμεσα στο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό φορέα. Φυσικά αυτό που χρειάζεται και ο δημόσιος και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις ε, είναι ένα ε, ανταγωνιστικό περιβάλλον με ισότιμους όρους όπου οι συμβάσεις ε, υλοποιούνται, υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός διευθέτησης διαφορών, αλλά είναι και ξεκάθαρο το φορολογικό σύστημα. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ είναι η ασφάλεια. Να υπάρχει ασφάλεια στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και θα, στο οποίο θα παράσουν τις υπηρεσίες τους. Χρειάζεται φυσικά επίσης ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν φραγμοί για τις ε, εξωτερικές επενδύσεις όπου μπορούν να επαναπατρίσουν τα μερίσματά τους απρόσκοπτα, όπου μπορούν να αποζημιωθούν, να ακόμη και αν διακοπεί ένα πρόγραμμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ρόλος της ΕΤΕ. Ποιος ε, ήταν, ε, λοιπόν, υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία ε, για τις δίτες στην ΕΤΕ, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός. Πέρυσι η ΕΤΕ χρηματοδότησε 16 προγράμματα για περίπου 3,5 δις ευρώ. Το προηγούμενο έτος ε, λίγο χαμηλότερο, 6 προγράμματα, αλλά γενικότερα κατά μέσο όρο 10 προγράμματα ΣΔΙΤ χρηματοδοτούνται από εμά το χρόνο κυρίως στον ενεργειακό τομέα, το τομέα της ίδρευσης ε, και των μεταφορών. Αυτοί οι τρεις τομείς Πιστεύω ε, καταλαμβάνουν και τις υψηλότερες θέσεις, ε, μάλλον τονίζονται ε, και στο έγγραφο εργασίας. Πρέπει να σας πω δε ότι για, σε πολλά από τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε υποστηρίζουμε τους Ευρωπαίους επενδυτές αλλά όχι μόνο, υποστηρίζουμε και τους σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, στο, στην Βόρεια ε, Κένια ε, χρηματοδοτήσαμε ένα αιωλικό πάρκο και είμαστε ένα από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες δεν χρειάζεται τώρα, δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειε για να εξηγήσω ακριβώς, τέλος πάντων, χρησιμοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και την εντολή κοτονού που έχουμε για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε εκεί και ε, υποστηρίξαμε το Βέστας που έδωσε τον εξοπλισμό, ε, τη Siemens και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα πλαίσια του προγράμματος υποστηρίξαμε πολλές εταιρείες και έτσι ε, θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να υποφεληθούν και να ανατεθούν οι συμβάσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Από πλευρά ΕΤΕ υποστηρίζουμε γενικότερα τους στόχους των πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάντι υποστηρίζουμε τα προγράμματα, ε, δίνουμε και τεχνική αρρωγή στις κυβερνήσεις αν χρειαστεί για να ε, συνάψουν οι ίδιες ΔΙΤ για τη στήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Επίσης, φροντίζουμε ώστε από τεχνικής, οικονομικής και νομικής άποψης να είναι τα προγράμματα ικανοποιητικά και στον τομέα των δημοσίων προμηθειών επίσης δραστηριοποιούμαστε και ε, ε, έχουμε και το, τη, τη μόχλευση διότι μπορούμε να δανειζόμαστε πολύ φθηνά και δίνουμε με πολύ παρατηταμένη περίοδο ρήμανσης ε, πολύ καλά δάνεια στις εταιρείες 15-20 χρόνια ή ακόμη και μεγαλύτερες περιόδους προβλέπουμε στους διαγωνισμούς και επίσης συνδυάζουμε τα δάνειά μας ε, και με ε, επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παραδείγματος χάρη, Υπήρξε ένα χρηματοδοτικό κενό στο πρόγραμμα που προανέφερα και χρησιμοποιήσαμε το equity stake Δηλαδή, ε, χρηματοδοτούμε εμείς και στη συνέχεια τα κονδύλια που δίνουμε χρησιμοποιούνται για άλλες ε, ε, αναπτυξιακές δράσεις. Να πω και κάτι τελευταίο για τις μεσογειακές χώρες και για τη Μέση Ανατολή έχουμε συγκεκριμένη προετοιμασία ανά των προγραμμάτων Το NET 5P χρησιμοποιείται χρηματοδότηση από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές το ποσό ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ ε, είμαστε βασικός εταίρος, ε, αλλά συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς όπως ε, η EBRD με την Αναπτυξιακή Υπηρεσία της Γαλλίας και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ολοκληρώνοντας να πω πως αυτό που χρειάζονται οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει είναι κατάργηση των φραγμών για τι εξωτερικέ επενδύσει όπω έλεγχο συναλλαγματικών ισοτιμιών, ε, παρεμπόδιση τη ροή των ε, μερισμάτων, ε, μια συνεπή και σταθερή φορολογική πολιτική, Για να προωθήσουμε αυτές τις αλλαγές από πλευρά ΕΤΕ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε σε πρόωρο στάδιο της κυβερνήσεως ώστε να ε, δημιουργήσουν αυτό το κατάλληλο το ε, πρόσφορο περιβάλλον για τις ΣΔΙΤ να ενισχύσουν το ε, ρυθμιστικό τους πλαίσιο, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ούτως ώστε να συναθούν ΣΔΙΤ. Δεν είναι πάντοτε εύκολο το έργο μας, ε, διότι ένα και περισσότερες χώρες, όπως ξέρετε, προσφεύγουν, μάλλον επιμένουν να υπάρχει ένα, ε, μια τοπική διάσταση όταν ε, συμμετέχουν σε διαγωνισμό για μια ανάθεση και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στην Νότια Αφρική, παραδείγματο χάρη, η κυβέρνηση ανέλαβε να προωθούσε ένα πρόγραμμα, τεράστιο πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κάθε στάδιο ε, ε, αυξάναν τις ε, απαιτήσεις που είχαν για την τοπική, το τοπικό κομμάτι των δραστηριοτήτων των εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Αυτό μας δυσκολεύει εμάς, διότι θέλουμε οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση για τις επενδύσεις τους και να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Από πλευράς μας λοιπόν σε μόνιμη βάση αυτό ε, επιχειρούμε στις σχέσεις μας με τις επιχειρήσεις. Όμως τις δείτε, βλέπουμε ότι ε, αυξάνεται αυτή η πρακτική και αυτό μας εμποδίσει. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κατά τα άλλα ε, οικονομικά βιώσιμα και υγιή προγράμματα. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ και αν έχετε δικό να ρωτήσετε, εδώ είμαι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσίες σας. Θα τις δούμε και στην αυθεντική τους μορφή. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για μια πολύ εστιασμένη και σύντομη τοποθέτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα για το σημαντικό αυτό θέμα. Έχουν εμπειρία. Τα κράτη από τις ρυθμίσεις αυτές που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές γιατί σε περιπτώσεις ε, ελλειπών δημόσιων πόρων μπορούν να αποτελέσουν αυτά τα κονδύλια και η διαχείριση σημαντικό καταλήτη για τις επενδύσεις και των υποδομών. Είναι πολύ ανταγωνιστικέ ήδη οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για ΣΔΙΤ σε όλο τον κόσμο. ΣΔΙΤ που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικέ επιχειρησιακές ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Όλο και περισσότερο όμως αναπτύσσεται και ο πολύ σκληρός ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε πολύ, πολύ προστατευμένες αγορές. Επομένως πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να δρουν σε μια προστατευμένη και ταγωνιστική αγορά οι επιχειρήσεις μας ώστε να περιορίσετε το κόστος. Για, αυτά τα, για αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε πρόσβαση χωρίς διακρίσεις για τις ΔΙΤ και συμμετοχή τους στις διεθνείς συναλλαγές για κρατικές επενδύσεις. Επίσης, με έμφαση τις επενδύσεις, η ΣΔΙΤ είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε σημαντικές ε, συνεργατικές σχέσεις, γιατί μπορούμε να διαπραγματευτούμε και δεσμεύσει για πρόσβαση στην αγορά για τις επενδύσει αλλά και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν, να διαδραματίσουν επιχειρήσεις σε τρίτε αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη ηγητέ, Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σε αυτή την πρώτη απόψη Να ευχαριστήσω βέβαια τον εισηγητή. για την έγγραφο εργασία, το οποίο είναι ευρύτατο και μας επιτρέπει να διαρευνήσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο το ζήτημα με την εξαιρετική βιογραφία που μας έχει προσφέρει. Έχω τις εξής παρατηρήσεις. Καταρχάς τον ορισμό της ΣΔΙΤ. Εμείς είμαστε υπέρ ενός ορισμού διεθνώς που να περιλαμβάνει και την παροχή των υπηρεσιών και την εξασφάλιση, την κατασκευή των υποδομών αλλά και να συμπεριλαμβάνει τους ε, ιδιώτες εταίρους για την κατασκευή του έργου χωρίς να περνάμε από ιδιωτικοποίηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία εταιρική σχέση ισοδύναμη, ισότιμη. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν ε, σε ορισμένε περιπτώσεις αναφερθεί και γραφτεί μπορούν να αποτελέσουν μια καλή εκκίνηση και να βοηθήσουν σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών για τις επενδύσεις, πρόσβαση στις αγορές, συμφωνίες με τέτοιες χώρες ή ομάδες τρίτων χωρών. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν μεγάλη τεχνογνωσία και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε περισσότερες αγορές. Και επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι έχει τεράστια σημασία να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα για το άνοιγμα των αγορών στα θέματα των δημοσίων αγορών, των δημοσίων συμβάσεων. Ιδιαίτερος δε εμείς, ως ΕΛΚΑ, υπερασπιζόμαστε αυτή τη δυνατότητα που αποτελεί ένα από τους κύριους πυλώνες. Έχουμε θετική αμοιβαιότητα ώστε να μην κλείνουμε την αγορά μας, αυτούς που κλείνουν τη δική τους και ταυτόχρονα μπορούμε να μιλήσουμε για όλες τις αγορές, δημόσιες αγορές, επενδύσεις για τις δημόσιες συμβάσεις που αποτελούν στη τελευταία ανάλυση και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, ασφάλεια, δικαίου, ασφαλές περιβάλλον για τις ΔΙΤ. Και άρα πιστεύω ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας μπορεί να προαγάγει την, ένα θετικό κλίμα για τις ΔΙΤ και να αποτελέσει υπό αυτή τη έννοια ένα καλό βήμα προόδου για τις επενδύσεις. θα ενθαρρύνουμε έτσι τις εταιρικές σχέσεις, ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την δημιουργία ενός κλίματος οικονομικού για τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητε τους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω και εγώ συγχαίροντας τον εισηγητή για το έγγραφό του Συμφωνώ με αυτό που προλαλεί σα και τα συγχαρητήριά του και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να χαιρετήσω τη συμβολή της και την εμπειρία της και να την ευχαριστήσω για τη δουλειά της. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι ΣΔΙΤ λόγω της μεγάλης αύξησή τους τα τελευταία χρόνια. Εγώ ήμουν υπεύθυνη στο Υπουργείο στην χώρα μου για τρία χρόνια περίπου για τις υποδομές επίγειων μεταφορών. Έζησα ακριβώς τις αλλαγές που είχαμε στην παροχή της υπηρεσίας μετά από τις ΔΙΤ και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ας πούμε το πώς θα μπορούσαμε μελλοντικά να βελτιώσουμε ιδιαίτερα στις τρίτες χώρες την αποτελεσματικότητά τους. Να πω πάντως ότι κυρίως μάλλον δεν είναι πάντοτε τα ΔΙΤ η καλύτερη απάντηση για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τιμής και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό και πιο σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή των προγραμμάτων χρηματοδότησης ώστε τα ΣΔΙΤ να συμφέρουν, να συνεισφέρουν αποφασιστικά. Αν τα, θε, τα θεωρήσουμε ως εργαλείο μείωσης δημοσίου χρέους, αυτό είναι λάθος. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε υποδομές ως υπηρεσίες που θα είναι πολύ δαπανηρέ, όχι μόνο για τους τωρινού πολίτες, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Θεωρώ εξάλλου ότι είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε τους κινδύνους. Γίνεται αναφορά στο έγγραφο αυτό. Κίνδυνο δημιουργίας υποδομών και μετά προσφορά και ζήτηση. Εγώ νομίζω ότι όπου υποχωρεί η ζήτηση, εκεί ακριβώς υποχωρούν και επιχειρήσεις και καταλήγουμε σε προσφυγές κατά της δημόσιας διοίκησης που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του έργου. Θα πρέπει λοιπόν οι κίνδυνοι να προσδιοριστούν σωστά ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του κινδύνου που πρέπει να αναλάβει ο ιδιωτικό τομέα και των εγγυήσεων που παρέχει η δημόσια διοίκηση. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η υπεύθυνη διαχείριση και οι υπηρεσίες που παρέχονται να διαθέτουν τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους ώστε να γίνεται ένα σωστό σχεδιασμός των ΣΔΙΤ να γίνεται επίσης σωστή παρακολούθηση της παροχής των υπηρεσιών και κυρίως να υπάρχει ένα σύστημα με δείκτες που θα επιτρέπουν στους πολίτες να παρακολουθούν και να επιβάλλουν κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν τις προσδοκόμενες υπηρεσίες. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να προωθήσουμε τα ΣΔΙΤ σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες προσδοκίες ανάπτυξης και όπου έχουμε συνάψει σημαντικές διεθνεί συμφωνίε. Θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να αναζητήσουμε την συνοχή μεταξύ αυτών που εμεί ασπιζόμαστε ω αρχή της δραστηριότητα και της επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής ευθύνη των επιχειρήσεων μα ώστε να τηρήσουμε αυτές τι αρχέ. Και τέλο, για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες να συμμετάσχουν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Στα μεγάλα προγράμματα χρειάζεται όγκος χρηματοδότης στον οποίο οι μικρομεσαίες δεν έχουν πρόσβαση. Είτε λοιπόν θα προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων και μικρών ή μεγάλων και μεσαίων ώστε να αποτελέσουν μαζί τμήμα των ΣΔΙΤ ή αυτό το σύστημα θα έχει δύσκολη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες. Κατά 95% λοιπόν έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, οπότε πρέπει να αναζητήσουμε συστήματα χρηματοδότησης και εργαλεία μέσω συμφωνιών συνεργασίας ώστε να υπάρχουν ομάδες που θα κάνουν προγράμματα επενδύσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, να σας πω ότι κατά την άποψή μας οι σοσιαλιστές θεωρούμε ότι τα ΣΤΙΤ δεν αποτελούν ιδιωτικοποίηση των κερδών που αντιστοιχούν στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας. Οι κίνδυνοι δεν αναλαμβάνονται από τα δημόσια ταμεία. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε ότι αποτελεί μια από τις βασικές μας αρχές και ότι δεν γίνεται να ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη και να κάνουμε δημόσια τα χρέη. Οπότε ώστε να πω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα προγράμματα ανάπτυξη εκτό συνόρων μα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το εργαλείο αυτό, ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξή του στι τρίτε χώρε και να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε. ώστε να υπάρχει και σωστή υπηρεσία μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίε και των δημοσίων αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σολάντσοβα, εκ μέρου των Φιλελευθέρων, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά. Ζητώντα συγγνώμη ότι θα πρέπει να φύγω αμέσω μετά, τη συνεδρία, αμέσως μετά την ομιλία μου, γιατί έχω και συντονιστέ στην εταιρεία. Ισδίτ. για να γυρίσουμε στο είναι πολύ σημαντικές και πηγή ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στην αναπτυξιακή μας συνεργασία μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά οι επιχειρήσεις μας μέσω των ΣΔΙΤ. Έχουμε ισχυρούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις και τις παραχωρήσεις έργων που αφορούν όλες ΣΔΙΤ. Πρόκειται για αρμοδιότητα τη Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς για κανόνες που ισχύουν, σα διαβεβαιώ, και εφαρμόζονται. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην επέκταση των κανόνων πέραν των συνόρων και τις βέλτιστες πρακτικές. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση στις ξένες δίτ. Δεν πρέπει να επιτρέπονται προς κόμματα διοικητικά ή άλλα. Και χρειάζεται να προστατευτούν οι επενδύσεις των επιχειρησών μας. στη χώρο της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας μπορούν να αξιοποιούνται μέσω των ΣΔΙΤ ποσά ε, ευρωπαϊκά ταυτόχρονα υποστηρίζοντας τις πολιτικές μας και οι ΣΔΙΤ θα είναι συμπληρωματικές βέβαια ως προς τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, τρέποντας ταυτόχρονα την καλύτερη αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Επίσης, θα ήταν καλή ευκαιρία της αξιολόγησης των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών και πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στον χώρο των ΣΔΙΤ, εφόσον δεν έχουν αντιμετωπιστεί κάποια προσκόμματα Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Φιέλνερ, ένα λεπτό μόνο. Μα νομίζω ότι το εξηγεί πολύ καλά ο εισηγητής τι σημαντικό πράγμα που είναι τα ΣΔΙΤ. Πολύ σημαντικές δε για την ανάπτυξη και κυρίως ε, στην ενέργεια και στον τομέα της ενέργεια και των υδάτων. Η ΕΤΕΠ ήταν νομίζω σαφέστατη στην ε, τοποθέτησή της και την έμφαση που έδωσε στη σημασία των ΣΔΙΤ για διμερείς ε, συμβάσεις και τη ρυθμίση, τη θέτηση διαφορών. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας όταν έχει να επεξεργαστεί θέματα επενδύσεων ε, και διθέτησης διαφορών για επενδύσεις. Να το θυμάται αυτό, δεν μπορούμε να λέμε από τη μια είναι σημαντικές οι και από την άλλη δεν θέλουμε προστασία των επενδύσεων η ρύθμιση, η διευθέτηση διαφορών. Θα ήταν υποκριτικό κάτι τέτοιο για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα η ΕΤΕΠ και αν δεν έχει χρόνο μας απαντήσει γραπτός να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στο ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις από ό,τι φαίνεται όπου απαιτείται η ύπαρξη διμερών συμβάσεων με μηχανισμούς διαθέτησης διαφορών ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντικές οι ΣΔΙΤ. Και άρα είναι καλό και απαραίτητο και εμείς να γνωρίζουμε ιδιαίτερα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν ε, τις επενδύσεις και τη διαθέτηση διαφορών για την ΕΤΕΠ. Τι σημαίνει επίσης έχει αυτό στις επενδύσεις ΕΤΕΠ. Και επίση πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να αποκλειστούν οι υπηρεσίες για το νερό, την ενέργεια από τη διευθέτηση των διαφορών ή την προστασία των επενδύσεων. Τι θα συνέβαινε αν ακολουθούσε τη γραμμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δυνατότητε θα είχε η ΕΤΕΠ να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα σημαντικά έργα που προάγουν την ανάπτυξη, την ενέργεια, τα ύδατα και την πρόσβαση σε αυτά σε όλο τον κόσμο ο πρόεδρος. Δύναμε να ζητήσω ακόμα τρία λεπτά από τους διερμενείς, Παρακαλώ, ώστε να μπορέσω να ξαναδώσω το λόγο στην ΕΤΕΠ και την κυρία Κέρνικ, εάν θέλει, για ένα λεπτό να απαντήσει. Ναι, και ήταν η ερώτηση άμεση προς εσάς. Δεν νομίζω ότι εγώ θα έπρεπε να απαντήσω. Οι νομομαθείς ε, που δουλεύουν στην ΕΤΕ πρέπει να το κάνουν πάντως. Ε, μπορώ να σας πω ότι λειτουργούμε βάσει διαφόρων συμφωνιών στην ε, Αφρική. Έχουμε τη Συμφωνία Κοτονού, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ε, στο δικό μου επίπεδο, φυσικά βάσει συμφωνία Κοτονού υπάρχει υποχρέωση για τις κυβερνήσεις, για να είναι διαθέσιμες ισοτιμίες. Αυτό προβλέπεται. Πάντως, για τις διμερείς συμφωνίες δεν θα το έλεγα διότι το σημαντικό είναι η δέσμευση που αναλαμβάνουν σε επίπεδο project, ε, σε επίπεδο εγγράφων ε, project για τις αγορές, για τις ε, προμήθειες, τι συμφωνεί από τη μία πλευρά δημόσιες φορές και από την άλλη επιχείρηση. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούνε οι νομικοί μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ας ακούσουμε τον εισηγητή μας. Θα το κλείσουμε. Πολύ χαίρομαι που σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Πολύ καλό είναι που δεν αγνοείται αυτό το διαθέσιμο εργαλείο. Μόνο, μόνο άρχισε η συζήτηση σήμερα, θα συνεχιστεί και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε, λέει ο Πράτος, έτσι και το σημείο 17. Το δω, σημείο 18. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλος ιδιαίτερος, διότι έγιναν πολλές παρουσιάσεις. Μετά θέλω να ε, ζητήσω συγγνώμη, διότι θα χρειαστεί να αναβληθεί η συζήτηση του σημείου 18. Είναι προφανές ότι γίνεται για λόγους περιορισμού, χρονικού περιορισμού. Να βάλε τη συζήτηση αυτό το σημείο για μελλοντική συνεδρίαση. τα διάφορα δεν νομίζω να υπάρχει τίποτε. 18 Μαρτίου θα γίνει, 18 και 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. τη συνεδρίαση.